Uh, colleagues, could we um, take our places? Thank you very much. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί που είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Χθε βέβαια είχαμε ακρόαση, μετά ξεκινήσαμε αμέσω την ε, συνεδρίασή μα Γι' αυτό θέλω να σα πω κάποια πρακτικά ζητήματα. Υπάρχουν τα πρακτικά τη 1ης και 2 η Ιουνίου στου φακέλου σα. Οπότε σα τα υποβάλλω προς έγκριση σήμερα. Αν έχετε παρατηρήσει, αντιρρήσει, να μα το έχετε πει παρακαλώ μέχρι αύριο το πρωί στι 12 το μεσημέρι. Αλλιώ θεωρούνται εγκεκριμένα. Δεύτερον, Θέλω να επενθυμίσω σε όλους σας ότι θα ψηφίσουμε στις 10 ακριβώς. Έχουμε μια μεγάλη ψηφοφορία του κυρίου Άρης Τζεβερία. Βέβαια πρώτα έχουμε να συζητήσουμε την έκθεση του κύριου Σβάμπ. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή μέχρι τις 10 θα ψεφίσουμε και μετά θα συνεχίσουμε. Επίσης, για μια απόφαση τώρα για εφαρμοστικά μέτρα όσον αφορά τα προϊόντα φώκιας. Η κυρία Βόλης ήταν χτες εδώ και είναι και υπεύθυνη από πλευρά τη Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Οπότε θα ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι την πρόταση που συζήτησε και οι συντονιστές χτες μετά την παρουσίαση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Αυτά για τα τυπικά. Οπότε ας ε, περάσουμε τώρα στη συζήτηση τη σημαντική έκθεση του κύριου Σβάμπ που είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι τα κεφάλαια 4 με 7 σήμερα. Έχουμε και τους σκιώδες εισηγητούς, την κυρία Κάπερ, τον κύριο Ρόσφορτ, τον Τιούνεν, ο κύριο Πίνα νομίζω δεν είναι εδώ, ο κύριος Τρενταφυλλίδης ναι, και ο κύριος Σαντίνη. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Θα δώσω το λόγο στον Ανδρέα Σβάμπ, ο οποίος μας ε, περιγράφει, μας έχει δώσει εδώ κάτι με γραφήματα έχρωμα που μας ε, εξηγεί κάπως την κατάσταση. Παρακαλώ κύριε Σβάπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. να παρουσιάσω τα κεφάλαια 4 και 5 και 6 αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχα μιλήσει για τα 1, 2 και 3, 2, 3 μαζί σημειωτέων. Προσπάθησα να τα παρουσιάσω με τρόπο κατανοητό όλα αυτά με κάποιες διαφάνειες χρήσιμες ελπίζω. Καλό είναι να συσκοτήσουμε λίγο την αίθουσα, να χαμηλώσουμε τα φώτα για να αρχίσουμε. Να πω καταρχήν ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έλαβα σχόλια και παρατηρήσεις, υποδείξεις από τους συναδέλφους, κυρίως από τους σκιώδες. Τα συμπεριέλαβα όλα αυτά και θα σας τα δείξω. Ως βάση συνολικά στο επίπεδο του ευρωπαϊκού δικαίου έχουμε 8 οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών και πολλές φορές λέμε, ρωτάμε γιατί ε, τις λέμε οδηγίες. Οι οδηγίες που αποτελούν τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου δεν πρέπει να συμπεριληφθούν μαζί. Κάποιες οδηγίες βέβαια είναι αλήθεια ότι ε, θίγουν επιμέρους τομείς, οπότε δεν μπορούν να συμπεριληφθούν. Αλλά οι τέσσερις οδηγίες που έχει ε, παρουσιάσει εδώ στους πυλώνες αυτούς οι Κομισιόν είναι αυτές που θα συνενωθούν και αντίθετα με αυτό που είπα στην πρώτη μου παρουσίαση όλες θα ενσωματωθούν στη νέα οδηγία. Γιατί το άλλαξα. Γιατί η κυρία Τούρνεν πολύ σωστά είπε ότι νομική περιπλοκότητα αν οι οδηγίες στα πλαίσια της ε, ελάχιστης εναρμόνισης παραμείνουν τότε θα αποτελεί πρόβλημα η νομική περιπλοκότητα και θα ήταν ιδιαίτερα σύνθετο οι ορισμοί στο κεφάλαιο 1 να περάσουν στις παλιές οδηγίες, γιατί θα έπρεπε να γίνει κάποια προσαρμογή. Άρα λοιπόν όλες οι οδηγίες που προτείνει η Κομισιόν να τροποποιηθούν θα περάσουν στην νέα οδηγία, οι παλιές θα καταργηθούν και έχουμε λοιπόν έτσι μία συνολική ρύθμιση για τις διατάξεις που προβλέπει η Κομισιόν. Στο κεφάλαιο 1 έχουμε ακόμα έναν τομέα ε, που περιλαμβάνει τις 8 οδηγίες για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που έχουμε κοινό ορισμό με το άρθρο 1 αλλά στο κεφάλαιο 2 και 3 το βλέπουμε με τη συνένωση αυτή, στο τέλος θα έχουμε κεφάλαιο 2, αυτό χρειάζεται. Γιατί χρησιμοποιήσαμε την αρχή της στοχευμένης, πλή, ε, της πλήρους εναρμόνισης και τα βγάλαμε τις ε, ε, πωλήσει ε, εκτός από που δεν γίνονται στην έδρα του πολιτή. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένες πωλήσει, σούπερ μάρκετ κλπ. που δεν εμπίπτουν εδώ. Ένα μεγάλο στοιχείο της συζήτησης βγαίνει με βάση την αρχή της πλήρους εναρμόνισης από το πεδίο εφαρμογής. Στα κεφάλαια 2 και 3 που παρουσίασα την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκα στους επιμέρους τομείς της πλήρους και ελάχιστης εναρμόνισης και γι' αυτό έχουν το χρώμα πράσινο-κόκκινο. Τώρα προστίθενται τα κεφάλαια 4 και 5 πάλι με χαρακτήρα κόκκινο-πράσινο και το κεφάλαιο 6 και θα μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες. Το κεφάλαιο 4 αφορούσε την προηγούμενη οδηγία για τα καταναλωτικά αγαθά εγώ προσπάθησα να ε, επιλέξω μια μέση οδό με την πρόταση που θα σας παρουσιάσω μια μέση οδό που δεν προσπαθεί να ε, επιτύχει συμβιβασμού στα τυφλά αλλά στοχευμένα να επιλέξει τομείς που ενδείκνυνται για μια συμφωνία όποια και αν είναι η μορφή της. Και γι' αυτό στο κεφάλαιο 4 έχω όλους τους κανόνες ε, που μπορούν να πλουστευθούν, να ε, γίνουν ενιαίοι δηλαδή, που είναι ο πράσινος τομέας στα πλαίσια της πλήρους εναρμόνισης ή τομείς όπου λόγω διαφορετικών συζητήσεων, δύσκολων συζητήσεων ε, δεν καταλήξαμε σε μία λύση και απόφαση. Εδώ μείναμε στην αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης και στο κείμενο η μορφή είναι εκείνη που προβλεπόταν στις παλιές οδηγίες. Άρα στο θέμα conformity, συμφωνία με τις συμβάσεις και το πέρασμα ή τη μεταβίβαση του κινδύνου από την, ε, πάμε από την ελάχιστη συμπλήρη εναρμόνιση, ενιαία, εις ό,τι αφορά το transfer of risk, μεταφορά κινδύνου, μέχρι τώρα σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη τους κανόνες της ελάχιστης εναρμόνισης τους είχαν εφαρμόσει. Μόνο στην Ιταλία από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μια διαφορά και εκεί μάλιστα ε, πάνε να καταργήσουν μια ασάφεια που επικρατεί. Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση κινδύνου, η, μετάβαση, η μεταφορά κινδύνου έχουν μια απλούστευση που ε, λαμβάνει υπόψη αυτό που αποτελεί κανόνα σήμερα. Σε ό,τι αφορά το τομέα του conformity, για το διασυνοριακό εμπόριο είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, έχω μείνει στην ε, πρόταση της Κομισιόν και λίγο έχω αλλάξει. Αυτοί είναι οι δύο τομείς στο κεφάλαιο 4 που θα πρέπει να ε, εναρμονιστούν στο 4, ιδιαίτερα στις εγγυήσεις και την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Στην, ε, έχουμε την ελάχιστη εναρμόνιση, δηλαδή την οδηγία των καταναλωτικών αγαθών που είναι στον κόκκινο, στο, με κόκκινο χρώμα. Ενδιάμεσα υπάρχει και ένας τομέας των προμηθειών των παραδόσεων, deliveries, και τα δικαιώματα εγγύσεων είναι με πράσινο-κόκκινο χρώμα οι δύο τομείς, αλλά ως επιτοπλίστων εντάσσονται στο, στην ελάχιστη εναρμόνιση. Σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις, μόνο η παράδοση ε, θα ε, αντιμετωπιστεί με νέο τρόπο στο μέλλον. Ό,τι δεν αφορά παραδόσεις δεν έχουμε εκεί εναρμόνιση. Εκεί τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στους ε, ισχύοντες κανόνες του στο εξεκουσιόν φορσέ του γαλλικού δικαίου, το αναθέτω εδώ ως παράδειγμα. Στον τομέα των δικαιωμάτων εγγυήσεων, το κείμενο της παλιάς οδηγίας ε, το συμπεριλάβαμε και εδώ και η παλιά οδηγία τότε είχε εναρμονίσει το, την επιλογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τώρα, η ιεράρχηση των δικαιωμάτων ποια θα είναι, αυτό εξακολουθεί να επαφίεται στα κράτη-μέλη και αναφέρομαι εδώ στην προηγούμενη οδηγία. Σε αυτό το τομέα, λίγο πολύ, ο τομέα του κειμένου της παλιάς οδηγίας συμπεριελήφθη, μόνο ο ορισμός της νέας, των νέων οδηγιών έχει προσαρμοστεί. Στο κεφάλαιο 4 βλέπετε καθαρά ότι πρόκειται για ένα συμβιβασμό μεταξύ του πράσινου κομματιού της εναρμόνισης και του κόκκινου που θα παραμείνει στα πλαίσια της ελάχιστης εναρμόνισης. Είναι όμως σημαντικό ότι και στον τομέα της ελάχιστης εναρμόνισης η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, ε, λήφθη ως βάση, είναι η απόφαση 64 του 2009, γιατί και το δικαστήριο λέει ότι στα πλαίσια της ελάχιστης εναρμόνισης είναι δυνατόν να ληφθούν από τα κράτη-μέλη αυστηρότερα μέτρα και τα μέτρα αυτά όμως θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εσωτερική αγορά θα λειτουργεί και για τους καταναλωτές και για τους επιχειρηματίες και γι' αυτό θα πρέπει να είναι αναλογικές, απαραίτητες οι διατάξεις αυτές για να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα κράτη-μέλη επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων τους να προβαίνουν σε αλλαγές, αλλά αν κάνουν αλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την αρχή που σας ανέφερα. Και στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών και Εσωτερικής Αγοράς αυτό είναι αυτονόητο. Πάμε στο κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 5... Αν πάρουμε ως μέτρο το πράσινο και το κόκκινο, ε, και εδώ βρίσκουμε μια συμβιβαστική μέση οδό, όμως είναι καθοριστικός ο τίτλος, ε, γιατί εδώ είναι μια σειρά απαγορευμένων ρητρών, δεν είναι η αναρμόνιση του μαύρου καταλόγου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα στο μαύρο αυτό κατάλογο να εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνουν όρους ε, που απαγορεύονται στην επικράτειά τους, όμως υπάρχει μία σειρά πω διατάξεις που προτείνομαι να εναρμονιστούν και υπάρχουν στο κείμενο. Υπάρχουν δηλαδή 5-6 ρήτρε που θα απαγορεύονται σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά ο κατάλογος είναι ανοιχτός και μπορούν τα κράτη-μέλη να προσθέτουν κι άλλες ρήτρε εάν το θεωρούν αυτό ενδεδειγμένο. Ε, στη συζήτηση ασκήθηκε ιδιαίτερη κριτική ότι ο κατάλογος αυτός θα ήταν ε, εξαντλητικός και είχε εναρμονιστεί. Όχι, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν την δυνατότητα να προσθέτουν ρήτρες που απαγορεύονται στην επικράτειά τους. ο γκρίζος κατάλογος που περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου είναι, ε, ε, υποτίθεται ή θα πρέπει να αποδειχθεί ο αθέμητος όρος. Εδώ υπάρχει ελάχιστη εναρμόνιση, αλλά στον τομέα του γκρίζου καταλόγου δεν θα ε, κάνουμε προτάσεις που θα ξεπερνούν τα όσα περιλαμβάνονταν στην παλιά οδηγία. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές εδώ, λίγος πολύ όπως το κεφάλαιο 4 ο κόκκινος τομέας περιλαμβάνει αυτά που ίσχυαν ήδη στην παλιά οδηγία στα πλαίσια της ελάχιστης εναρμόνισης. Αλλά και εδώ ισχύει η απόφαση που προανέφερα ότι τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να προσθέσουν νέες ρήτρες και να διατηρήσουν τις παλιές ρήτρες, όμως μόνο όταν οι νέες ρήτρες συνάδουν με την αρχή της, ελεύθε... της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό είναι και το ουσιαστικό νομικό κομμάτι του κεφάλαιου 5 και πάμε στο κεφάλαιο 6 που αναφέρεται λίγο και το 7 γιατί τα έχουμε συνδυάσει για να έχουμε μια εποπτεία καλή. Στο κεφάλαιο 6 και το αρχίσαμε να το λέμε αυτό στη χτεσινή συζήτηση Ορισμένα σημεία από την οδηγία για τις υπηρεσίες έχουν ε, υιοθετηθεί. Δεν ε, έχω την προσδοκία η διαδικασία peer review, αξιολόγηση κλπ. που προβλέπεται σε εκείνη την οδηγία να αποτελέσει πρότυπο, αλλά καλό θα ήταν και σε άλλα δύσκολα σημεία, σε άλλου δύσκολου τομεί τη ε, εναρμόνισης εσωτερική εσωτερικής αγοράς να τα κάνουμε αυτά, όπως την οδηγία για τις υπηρεσίες, ε, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 4, καλούμε τα κράτη-μέλη να ε, δηλώσουν τις τους διαφορετικούς εθνικούς κανόνες τους και να τους κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το μέτρο για την αιτιολόγηση της λογικής των εθνικών κανόνων θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητά τους και η χρησιμότητά τους για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένη χρησιμότητα, συγκεκριμένο όφελος, δηλαδή αφενός στις ε, συναλλαγές με τους επιχειρηματίες και το όφελος για τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά τη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών όταν πρόκειται για δικαστικές προσφυγές κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν να επιβάλλουν, να ασκούν τα δικαιώματά τους οι καταναλωτές αποτελεσματικά με όσο γίνεται λιγότερο κόστος και αυτό ε, προβλέπεται και στο peer review. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δηλώσουν γιατί είναι καλύτερο το δικό τους δίκαιο στο κεφάλαιο 4 για τους καταναλωτές από ό,τι τον, του γειτονικού κράτους και από τη συζήτηση αυτή θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και στοχευμένα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τι είναι σκόπιμο για τους καταναλωτές και όχι τι θα ήθελαν τα κράτη-μέλη και μόνο ή τι θα ήθελαν άλλοι stakeholders εμπλεκόμενοι. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 υπάρχει και μία δυνατότητα κάπως πιο έντονα σε σχέση με την προηγούμενη οδηγία οι εμπλεκόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι και οι καταναλωτικές οργανώσεις των καταναλωτών να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις τρευλώσεων, καταχρήσεων κλπ. Στο, ε, στα πλαίσια του δικαίου, των καταναλωτών να ενημερώνουν ε, και η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι στα πλαίσια της επιτροπολογίας αλλά με κανονιστική διαδικασία θα μπορεί να δημιουργεί απαγορεύσεις ρητρών στην εσωτερική αγορά. Και ε, όπως είπαμε στην αρχή η Κομισιόν καλείται την εξέλιξη αυτή στον τομέα ε, και πάνω στη βάση του, α, της απόφασης του δικαστηρίου που προανέφερα, ενδεχομένως να κάνει μια προσαρμογή και το, του δικαιικού συστήματο των κρατών μελών να το εξετάζει κάθε τρία χρόνια και να διαπιστώνει ότι πράγματι συμμορφώνεται προ την εσωτερική αγορά και τι αρχέ τη και να βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα για του καταναλωτέ αφενός αλλά και αφετέρου για του επιχειρηματίε στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά. Και με τι εκθέσει αυτέ, η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προτάσει και να τι ζητούμε και εμεί προτάσει. Το κεφάλαιο 6 λοιπόν ασχολείται με θέματα διαδικαστικά και γι' αυτό το, το κεφάλαιο 1 και 6 σημειώνονται με κίτρινο, δεν έχουν σχέση δηλαδή με την ε, πλήρη και ελάχιστη εναρμόνιση. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, ελπίζω ότι μπόρεσα να σας δώσω μια ε, ξεκάθαρη εικόνα για τις ε, προθέσεις μου σχετικά με την πρόταση που θα υποβάλω. Βεβαίως είναι δυνατόν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές για επιμέρους κράτη-μέλη. Βέβαια αυτή η οδηγία δεν θα ικανοποιήσει 100% τους πάντες. Αυτό νομίζω ότι το έδωσα να το καταλάβετε. Αλλά οι προτάσεις προέρχονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και γι' αυτό νομίζω ότι ο συμβεβασμός είναι αρκετά επιτυχημένος γιατί υπάρχει ένα δούνε και λαβίν αρκετά σημαντικό και αποτελεσματικό και ε, σε αυτό το σημείο περιμένω τα δικά σας εμπεριστατωμένα ε, σχόλια, τι ε, ανάγκες έχετε για αλλαγές κλπ. Για το χρονοδιάγραμμα να σας πω ότι το ενοποιημένο κείμενο είναι έτοιμο και το έχετε λόγω των μεταφραστικών διαδικασιών στο Κοινοβούλιο δεν, μπορούμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε το κείμενο στις δύο γλώσσες, δίγλωση μορφή. Σήμερα το απόγευμα θα το έχετε στα γερμανικά με το, την αιτιολογική έκθεση και μετά ενοποιημένο θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και θα έχουμε και το δίγλωσο κείμενο το οποίο με τις δύο στήλες, το οποίο ε, θα στηρίζεται στο ενοποιημένο, θα μεταφραστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα Ελπίζω να το έχουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Όλα τα έγγραφα πάντως σήμερα είναι διαθέσιμα και προτείνω να ε, ε, δώσουμε μια τρίμηνη περίοδο για επεξεργασία των τροπολογιών, οπότε στο τέλος Σεπτεμβρίου να είμαστε σε θέση να δούμε και να συζητήσουμε επί της ουσίας τις τροπολογίες. Γιατί αφενός πιστεύω ότι θα μπούμε στην ουσία όταν θα έχουμε μεταφρασμένες και όλες τις τροπολογίες και να μην μιλάμε μόνο πάνω στη βάση του δικού μου κειμένου και να μπούμε από εκεί σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεύτερον, σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή είναι πολύ δύσκολη η συζήτηση στο Συμβούλιο μετά την πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει και εμείς να επιδείξουμε κάποιο δυναμισμό στη συζήτηση, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να σπρώξουμε μπροστά τη διαδικασία. Και ο στόχος θα πρέπει να είναι μια συζήτηση τέλος Σεπτεμβρίου επί της ουσίας του περιεχομένου. Ε, θα την περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Σβάμπ, για τις λεπτομερείς εξηγήσει. Νομίζω ότι η διαφάνεια σας είναι πολύ πλήρης για τις προτάσεις που μιλήσαμε και ούτως ή άλλως ε, στις 12 Ιουλίου θα κάνουμε μια περαιτέρω συζήτηση για όλα τα κεφάλαια και ενδεχομένως Εκεί θα δούμε πώς όλα τα κομμάτια του, του συνδέονται μεταξύ τους. 13 Σεπτεμβρίου και μετά 29 Σεπτεμβρίου είναι οι επόμενες ε, εξετάσεις. Επομένως έχουμε χρόνο α, για να τα εξετάσουμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Θα σταματήσουμε στις 10 και αν ε, διεκπαιρεώσουμε γρήγορα την ψηφοφορία μπορούμε να επανέλθουμε. Καταρχάς, ε, η κυρία Γκέπχαρτ από τους Σοσιαλιστές έχει το λόγο. thank you, thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σβάμπ για την παρουσίαση. Έχω μπερδευτεί, για να σας το πω έτσι, ομά. Σε κάθε συνεδρίαση παίρνουμε και άλλο κείμενο, άλλη βάση. Σε κάθε συνεδρίαση μας δίνεται άλλη εποπτεία σχετικά με το πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα. Καταρχήν η ομπρέλα με τους τομείς, μετά η ομπρέλα χωρίς τους τομείς, μετά είχαμε μόνο τομείς. Ε, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο κύριε Σφάμπ και πρέπει να πω ότι πραγματικά έχω μπερδευτεί. Η μεσαία μηχανία. Γιατί δεν είναι διαφανής ο τρόπος εργασίας σας. Δεν φαίνεται που προς τα που πάτε. Θα επανέλθω σε αυτό. Καταρχήν κάποια σημεία ε, ουσίας θα αναφέρω και μετά θα παρουσιάσω το συνολικό, τη συνολική μου κρίση για να εκφράσω και τη δυσαρέσκειά μου. Θα δώσω τρία παραδείγματα, αν και θα μπορούσα να προσθέσω και πολλά περισσότερα. Πρώτο παράδειγμα, οι δυνατότητες του άρθρου 26. Λέτε ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής και ελάχιστη εναρμόνιση. Αλήθεια είναι αυτό. Όμως όταν συγκρίνω το κείμενό σας με αυτό της αρχικής οδηγίας, η δυνατότητα της επιλογής περιορίζεται πολύ για τα κράτη-μέλη. Περιορίζεται σε δύο δυνατότητες. Βελτίωση ή διορθωτικά μέτρα και αποζημίωση. Στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρεται σαφώς ότι υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η τρίτη καταργείται. Όχι, ο, ναι, και έτσι χειροτερεύει το βρετανικό δίκαιο. Γιατί στη στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενδιάμεσα, αν θα γίνει δηλαδή ε, μια διόρθωση, επιδιόρθωση των ελαττωματικών ή αν θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω ή αν θα μειωθεί η τιμή του προϊόντος, ενώ εσείς περιορίζεστε σε δύο δυνατότητες, α και β, ε, αποκατάσταση των, ή μείωση της τιμής. Δηλαδή η επαναχώρηση από την σύμβαση διαγράφεται από την πρότασή σας και αυτό χειροτερεύει την κατάσταση και σε σχέση με το δίκαιο που ίσχυε στην προηγούμενη οδηγία. Δεύτερο παράδειγμα. Επιδίνωση σε ό,τι αφορά το γερμανικό δίκαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις και τους όρους των συμβάσεων, των συμβατικών όρων που θα πρέπει να παρουσιαστούν. Εκεί χειροτερεύεται το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού λέτε σαφώς, μάλλον όπου λέει σαφώς ότι η δυνατότητα ανάγνωσης των συμβατικών όρων μπορεί να εξασφαλιστεί για τον καταναλωτή εφόσον οι συμβατικοί όροι και αυτό ε, θα, του δοθούν μετά από επιθυμία του. Αυτό το διαγράφεται την επιθυμία του. Οπότε λέει θα, θα είναι συνημένα. Άρα διαγράφεται τη δυνατότητα να επιτρέπεται ε, να δίνονται οι συμβατικοί όροι. Δηλαδή η σύμβαση θα συνοδεύεται από τους όρους της σύμβασης και μπορείτε να το διαβάσετε. Καμιά φορά ίσως ούτε και να κρατήσετε τους όρους αυτούς. Ε, το βίσκασε γιατί ε, το, το γαλλικό και αυτό το επιτρέπεται στο άρθρο 28 αναφέρεται αυτό και στο 42β στην αιτιολογική σκέψη. Ε, όμως ε, παίρνετε κάποια προϋπόθεση, μάλλον περιορίζεται το γαλλικό δίκαιο όπως ε, προβλέπετε και είναι δύσκολο να οριστεί τι είναι αυτό το εκ των όνου κάνευ, δηλαδή απολύτως, απολύτως απαραίτητο. Αυτό το απαραίτητο, unbedingt στα γερμανικά, δεν υπάρχει στα γαλλικά, άρα περιορίζεται το γαλλικό δίκαιο. Αυτά είναι τρία παραδείγματα τα οποία διάλεξα από το κείμενο που συνιστούν επιδίνωση. Ακόμα και αν έχουμε ελάχιστη εναρμόνιση επιδεινώνεται η βάση του δικαίου σε σχέση με, το αρχικό, με τα αρχικά κείμενα των οδηγιών. μπορείτε να ανέβετε αρνητικά όσο θέλετε, αλλά έτσι είναι όπως τα λέω γιατί εγώ το διάβασα και το ήλεγξα. Τώρα, το άλλο που θέλω να πω και τώρα παραπέμπω στο, στα γραφήματα και στις διαφάνειες, ε, που αναφερθήκατε στα κεφάλαια 1, 2, 3. Με τη νέα προσέγγιση σας προκύπτει πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ χειρότερο από αυτά που είπα μέχρι τώρα. Τα κεφάλαια 1, 2, 3 αρχικά τα είχατε στηρίξει σε ένα άλλο μοντέλο και είχατε διαγράψει πολλές διατάξεις από το κείμενο και είχατε πει ότι δεν θέλετε πλήρη εναρμόνιση αλλά θα μένατε στην ελάχιστη εναρμόνιση στις προηγούμενες οδηγίες. Αλλά αυτή την προσέγγιση την αλλάξατε. Δεν πήραμε καινούριο κείμενο για τα κεφάλαια 1, 2, 3. Οπότε όλοι οι τομείς που μέχρι τώρα καλύπτονταν από την ελάχιστη εναρμόνιση, τώρα δεν παρουσιάζονται, δεν περιλαμβάνονται στην καινούργια σας πρόταση. Άρα δεν βρίσκονται στα πλαίσια της ελάχιστης εναρμόνισης πια. Και αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά τα κράτη-μέλη τώρα μπορούν να εισάγουν χειρότερες διατάξεις από εκείνες που είχαν στα πλαίσια της ελάχιστης εναρμόνισης. Και αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Η ομάδα μου ποτέ δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση, γιατί αυτό σημαίνει σε απόλυτους όρους επιδείνωση του δικαίου για τους καταναλωτές. Το σκέφτηκα πολύ, γιατί δυσκολευόμουν να καταλάβω τι ακριβώς κάνετε, πώς προχωρείτε, τι στόχο έχετε θέσει. Η αδιαφάνεια της προσέγγισής σας τι σημαίνει. Νομίζω ότι σήμερα ε, βγάλατε λίγο τη μάσκα δεν σας ενδιαφέρει περισσότερη προστασία των καταναλωτών, αλλά η λιγότερη και θέλατε να το καλύψετε αυτό μέσα από την αδιαφάνεια. Αλλά δεν γίνεται. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει η ομάδα μου. Εγώ ήρθα και μάλιστα την Τρίτη όταν στην ομάδα εργασίας συζητήσαμε το θέμα είχα πει στους συναδέλφους μου ότι σήμερα ήθελα να ήμουν διπλωματική, να χρησιμοποιήσω διπλωματική γλώσσα. Αλλά δεν είχα δει το κείμενό σας, ούτε είχα δει τα σημερινά. Οπότε ε, έσπασα, παραβίασα την, την υπόσχεση που είχα δώσει, ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, αλλά εδώ πρέπει να μιλήσω με ξεκάθαρη γλώσσα και θα πρέπει βέβαια να σας πούμε τι μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε και τι δεν μπορούμε σε αυτή την οδό δεν θα σας ακολουθήσουμε. Οπότε θα κάνω αυτό που σκεφτόμουν να κάνω από την αρχή. Στις τροπολογίες που θα καταθέσω ως βάση θα πάρω το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι το δικό σας γιατί είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες τις οποίες εμείς με αυτόν τον τρόπο θα τις βάλουμε πάνω στο τραπέζι, θα τις συζητήσουμε και θα τις ψηφίσουμε. Αλλά αυτά εδώ που μας παρουσιάζεται είναι πολύ αδιαφανή και δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει πού αποσκοπείται και τι θα βγει στο τέλος. Η ομάδα μου δεν μπορεί να συμφωνήσει και τέλος να με, συμφω... να συγχωρείτε για την ξεκομμένη μου γλώσσα. Δεν είναι προσωπική επίθεση, είναι ε, καθαρά πολιτική θέση. Ε, εγώ και η ομάδα μου δεν μπορούμε να εργαστούμε με μεθόδους που δεν παραδεχόμαστε. Δεν θα τις ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ για τα πολύ ειλικρινή σας ε, σχόλια και είναι σημαντικό να διατυπώνονται αυτά τα σχόλια. Ως πρόεδρος θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση. Από αυτά που κατάλαβα, από αυτά που είπε ο εισηγητής, είμαστε σε θέση να έχουμε ένα πλήρες κείμενο που καλύπτει όλη την οδηγία και όλα τα τμήματα της οδηγίας. αναφερθήκαμε και σε κάποια σημεία που θα τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά βέβαια τον, τον Ιούλιο. Πάντως ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές καλό θα ήταν να βρεθούν λιγάκι μαζί με το κείμενο το ενιαίο ε, πριν συναντηθούμε στις 12, κάποια στιγμή στο Στρασβούργο, ούτως ώστε να, δούμε, να δείτε μάλλον που βρίσκεστε. Ο κύριος Χοσφόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ίσως με πιο διπλωματική γλώσσα από την Εύελιν, αλλά δεν είναι και δύσκολο να μιλήσω πιο διπλωματικά από την Εύελιν. Θα συμφωνήσετε όλοι. Αγαπητέ Ανδρέας, ε, Κάποιε από τι επικρίσει τη Εβελίν είναι βάσιμε, αλλά εγώ θεωρώ ότι βελτιώνεται το κείμενο σε σχέση με το κείμενο τη Κομι... Κομισιόν. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι απόλυτα ικανοποιητικό, αλλά θεωρώ ότι το βελτιώνεται. Α ξεκινήσω από τη φιλοσοφία, που είναι και σημαντικό πράγμα. Είστε λιγάκι μάγο, έτσι. Προσπαθείτε πέρα από το να βρείτε τη χρυσή τομή, να συμφιλιώσετε την, ενα... την ε, ελάχιστη εναρμόνιση με τη μέγιστη εναρμόνιση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ε, αν φτάσουμε, αν βρούμε τη χρυσή τομή ή μάλλον το μέσο όρο, ε, τελικά δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε η Εύελιν, μπορεί να είναι σωστό, ότι δεν καταλαβαίνουμε το σκοπό. Ειλικρινά σας λέω, αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ένωση, την χρηματοπιστωτική κρίση, την οικονομική κρίση, το γεγονός ότι λέμε ότι ενδεχομένως μερικές φορές υπάρχει μια δυνατότητα να έχουμε μια θεώρηση της Ευρώπης που ε, παντρεύει το στόχο ε, της ε, με τους εθνικούς στόχους δεν είναι άσχημη ιδέα. Ε, δεν είναι λύση για όλα τα προβλήματα, δεν είναι πανάκια, αλλά είναι ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχει ένα μη καινοτόμο στοιχείο το οποίο τονίζεται και που είναι η σπονδυλική στήλη του κειμένου που μας απασχολεί. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη ενέκριναν τις, και θα εγκρίνουν τις εξαιρέσεις που θα επιβάλλουν. Βασικά αυτό είναι ο ακρογωνιαίος αλήθος του κειμένου σας. Δηλαδή, οι εθνικές διατάξεις, ε, η ελάχιστη εναρμόνιση θα υπάρχουν, αλλά εφόσον υπάρχει απόδειξη, εφόσον μπορούν να δικαιολογήσουν αυτά τα μέτρα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε συνεχεία ε, κατά πόσο είναι αποτελεσματική αυτή η λύση. Αν δίνουμε απλώς ε, επιταγή λευκό στην ε, Κομισιόν για να κάνει ό,τι θέλει, δεν, δεν θα λειτουργήσει το πράγμα. Υπάρχουν δύο κριτήρια και στο κείμενό σας και προσθέσατε άλλο ένα στην, προσωπική, στην προχωρική σας παρέμβαση. Τα δύο που βάζετε στο κείμενο είναι ε, οι εμπορικές πρακτικές. Ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο τις ε, γλωσσικές μεταφράσεις ε, σε κάθε γλώσσα. Σήμερα είπατε σύγκληση στην ενιαία αγορά. Δεν το λέτε έτσι στο κείμενο, αλλά με αυτό το στόχο συμφωνούμε όλοι. Αλλά λέτε επίσης απόδειξη και στις διάφορες ε, δικαστικές διαδικασίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Πρέπει να δούμε το δίκαιο από χώρα σε χώρα. Και εγώ φυσικά δεν είμαι νομομαθής. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η υπεράσπιση του καταναλωτή. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ. Τι θα συμβεί στην περίπτωση όπου για διάφορους λόγους στα διάφορα κράτη-μέλη τα δικαστήρια δεν εξέτασαν την υπόθεση των καταναλωτών, είτε γιατί οι καταναλωτές δεν προσέφηγαν σε αυτά, είτε γιατί δεν μπορούν να προσφύγουν. Σε αυτή την περίπτωση ανακαλείται ή, αυτή είναι η μία μια ή αν δεν υπάρχει δικαστική διαιτησία, δεν είναι αυτό κριτήριο για την απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να το διερευνήσουμε αυτό το σημείο. Υπάρχει ένα καινούριο ε, εργαλείο ενδιαφέρον. Εν συνεχεία, είμαστε ουσιαστικά κάπου ε, πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Θα πρέπει να δούμε από πού θα πέσουμε, από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε ένα κεντρό κόμμα, μια κεντρό απαράταξη. Σίγουρα ε, στις εγγυήσει ε, του συμβολέου ε, θα πρέπει να μπουν και τα εξαρτήματα. Αυτό είναι βελτίωση. Αυτό που λέτε ότι η κακή εγκατάσταση ενός αγαθού είναι ένα ελάττωμα όταν αυτό υπάρχει στη σύμβαση και αυτό είναι πρόοδος. Η δυνατότητα προσφυγής του καταναλωτή ε, υπό τον όρο ότι είναι εύλογο και όχι δυσανάλογο ε, αυτό το μέτρο και αυτό είναι χρήσιμο. Ε, κάτι άλλο. Σε μια πρόσφατη συνεδρίαση ε, παρενέβην και είπα υπάρχει το εξής δικαίωμα. Μερικές φορές θα πρέπει να διακρίνουμε τον τελικό έμπορο από την προηγούμενη αλυσίδα. Ε, αυτό είναι θετικό που το ξαναβάζετε στο κείμενο για τη δυναμική της εσωτερικής αγοράς. Φυσικά υπάρχουν ερωτήματα για το άρθρο 26. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Εύελιν. Με μία μικρή απόχρωση όμως διαφορά. Δηλαδή διατηρείται τη δυνατότητα ε, λύσης του συμβολέου, αλλά το βάζετε ως δευτερεύον στοιχείο. Δηλαδή δεν είναι πρωτεύον στοιχείο. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα απόρριψης βρετανικό δίκαιο υπάρχει θα πρέπει, και αυτό θα πρέπει να μπει στην περίπτωση των εξαιρέσεων που επανισάγουν τα κράτη. Αλλά δεν υπάρχει ε, ως γενικό στοιχείο. Εγώ θα ήθελα να, να υπάρχει ως γενική δυνατότητα. Εσείς δεν το προτείνετε για την βελτίωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Καλό θα ήταν να το συζητήσουμε. Έχω και άλλα στοιχεία την εισαγωγή ενός, μιας επιπλέον προθεσμίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σεβασμός της προθεσμίας παράδοσης. Αυτό νομίζω ότι μειώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών στη Γαλλία. Γιατί στη Γαλλία θεωρητικά, ακόμη και αν δεν εφαρμόζεται καλά, όταν δεν σεβόμαστε το, την προθεσμία αυτή, υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης του συμβολέου. Υπάρχει και μια δεύτερη προθεσμία, την οποία βάζεται, θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Ε, υπάρχει κάτι που βάζεται ως βελτίωση. Το γεγονός ότι ο, ο μπορεί ο ίδιος να επανορθώσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και να του επιστραφούν τα χρήματά του από τον έμπορο. Φυσικά εσείς λέτε ότι τα έξοδα αυτά θα πρέπει να είναι εύλογα. Αλλά πώς θα υπάρξει συμφωνία πριν από την επιδιόρθωση. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Δεν συμφωνώ για το σημείο που αποκλείουμε τις εξατομικευμένες ε, ρήτρε ε, του πεδίου του άρθρου 30. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες μερικές φορές οι καταναλωτές να πέσουν θύματα. Γιατί αν αρκεί να προσθέσουμε μία επιπλέον φράση σε, μια, σε ένα κλασικό συμβόλαιο και να πούμε ότι δεν είναι κλασικό συμβόλαιο, αλλά ε, είναι ένα συμβόλαιο στο οποίο παρεμβαίνει ο καταναλωτή και να το αποσύρουμε από αυτό το συμβόλαιο τη δυνατότητα εφαρμογή τη συμβατική ρήτρα. αυτό είναι συζητήσιμο. Δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι. πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν. Όπω είπατε τώρα, χρειαζόμαστε τρει μήνε για να βρούμε συμβιβασμού. Ελπίζω να πάμε μακριά. Έχουμε ένα μείζωνα στόχο να μην υποβαθμίσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να πάμε στι πατρίδε μα και να πούμε στου καταναλωτέ μα μειώνουμε τα δικαιώματά σα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα μία ένα, έτσι, ένα ρηθέν. Ε, σας παραπέμπω στο, στο ποδο, όχι στο ποδόσφαιρο, αλλά στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Ε, κύριε Ανδρέας, είσαστε καλός πατινέρ. Υπάρχουν οι ελεύθερες ασκήσεις και οι επιβεβλημένες στις επιβεβλημένες. Θα πρέπει να, το, να κάνουμε τις επιβεβλημένες ασκήσεις για να φτάσουμε στην ε, μέγιστη εναρμόνιση. Ορισμένα πράγματα είναι ε, επιβεβλημένα ε, και για το πνεύμα της οδηγίας, αλλά και για τη βελτίωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Και έπειτα, οι ελεύθερες ασκήσεις. θα πάρουμε λίγα ρίσκα, θα κάνουμε προσπάθειες. μερικές φορές υπάρχουν κίνδυνοι, μπορούμε να στάσουμε τα μούτρα μας, αλλά για να τα καταφέρουμε θα πρέπει να πάμε καλά και στις ελεύθερε ασκήσεις και, σε, και στις υποχρεωτικές ασκήσεις. Αυτά και δεν έκανα την κλασική, το κλασικό αστιάκι με το ποδόσφαιρο, παρότι είναι πολύ επίκαιρο. Σίγουρα με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, σφιχτό χρονοδιάγραμμα και πρέπει να προχωράμε γρήγορα. Σίγουρα ο κύριος Σβάμπ θα μπορέσει να προχωρήσει στη ζήτηση σε λεπτομέρειες. Σίγουρα θα το συζητήσετε ε, κι εσείς ε, με τον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, για κύριε Λάντεν. Θέλω πρώτα απ' όλα η κυρία Λόκεγκάρτ. Να σας πω πως είναι ένα περίπλοκο θέμα, ιδιαίτερα ευρύ. Είναι τιτάνιο το έργο μας. Για τον εισηγητή και για τους σκιώδεις εισηγητής, οι εισηγητές αυτό που ισχύει είναι ότι πρέπει να μελετήσουν όλα τα άρθρα, άρθρο προς άρθρο, να δούνε τι είναι λογικό, τι δεν είναι, να διασταυρώνουν κάθε τόσο τα όσα αναφέρονται στο κείμενο για να βλέπουν κατά πόσο στέκουν. Έτσι κι αλλιώς Είμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που συμμερίζετε την, ε, τις επικρίσεις μας για την κατανομή. Είναι θετικό αυτό. Εκεί που έχω όμως κάποιες αμφιβολίες είναι όσον αφορά το καθεστώς, όπως έλεγε και Ευλήν, των κεφαλαίων 1, 2 και 3. Ίσως πρέπει να διατυπωθούν εκ νέου, γιατί έχουμε βγάλει ένα τόσο μεγάλο μέρος του κειμένου που τελικά δεν ξέρουμε αν πρέπει να διατηρήσουμε την οδηγία ή όχι. Μήπως πρέπει να την εγκαταλείψουμε εντελώ. Πρέπει να ξαναδούμε το κείμενο δηλαδή. Τη διατύπωση. Χρειαζόμαστε ένα συνολικό κείμενο, παγιωμένο. Για τους σκιώδες εισηγητές είναι σημαντικό αυτό. Έτσι κι αλλιώ έχουμε και διακοπές, άρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακριβώ τρει μήνες στη διάθεσή μας για να δουλέψουμε. Η συζήτηση, λοιπόν, επί τη ουσία πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ας πούμε 20 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον για να έχουμε χρόνο να δουλέψουμε σωστά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, για τα κεφάλαια που μας παρουσιάσατε σήμερα. Υπάρχουν βελτιώσεις, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά όπως έλεγε και ο κύριος Ροσφόρ, υπάρχουν και σημεία που επιδεινώνονται. Μιλάτε για ένα μέσο όρο, για μια μέση οδό. Δεν είναι όμως εύκολο. Η βασική αρχή έχει ήδη καθοριστεί. Το είπαμε από την αρχή, είναι το άρθρο 4. Θέλουμε να καθορίσουμε μια βάση πλήρους εναρμόνισης με εξαιρέσεις. Ή αλλιώ ας πούμε ότι ξεκινάμε από το ελάχιστο και σε άλλα σημεία να λέμε ποιο είναι το ανώτατο. Μα δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση σήμερα. Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου θα πρέπει να ορίζουμε τι σημαίνει εναρμόνιση για το κάθε κεφάλαιο. Ποια είναι τα άρθρα για το οποίο έχουμε πλήρη εναρμόνιση. Για μένα μια τέτοια προσέγγιση είναι προτιμότερη. Έρχομαι τώρα στο κεφάλαιο 4 και θα πάω γρήγορα κύριε Χάρμπορ, ναι. Κεφάλαιο 4 λοιπόν. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια και τα ίδια. Η επιπλέον προθεσμία των 7 ημερών δεν είναι πάντα υπέρ του καταναλωτή, γιατί περνάμε από 30 σε 37 μέρες για να καταγγελθεί συμβόλαιο. Άρθρο 24. Πλήρης εναρμόνιση. Μα εδώ πρέπει να σκεφτούμε πολύ τα πράγματα και την, να δούμε την εθνική νομοθεσία κάθε φορά για να δούμε Να δούμε κατά πόσο λοιπόν η πλήρη αναρμόνιση εδώ είναι η σωστή λύση όχι. Είναι κάπως επικίνδυνο. 6. Αναφέρθηκαν σε αυτό και η Ευλίν και ο κύριος Ροσφόρ. Είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν περισσότερα. Είναι αυτή η μεσιοδόση στην οποία αναφέρθηκα πριν. Και αυτό όμως αν υπάρχει κάποια αναλογία και αν είναι αποτελεσματικό το αυτό που θα γίνει. Ποιος όμως θα αποφασίσει για την αναλογικότητα ή για την αποτελεσματικότητα. Ποια είναι τα κριτήρια. Ποιος θα το αποφασίσει αυτός. αυτό για να πει ότι είναι αποτελεσματικό το μέτρο ή αναλογικό. Ποιος θα σας το πει αυτό αν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή. Εδώ δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Θέλω να ξέρω οι νομικοί στα διάφορα κράτη-μέλη τι θα πούνε. Θα τραβάνε τα μαλλιά τους. Γιατί δεν θα βγάζουν άκρη. Πώς θα ξέρουν. Αυτά, αυτό με απασχολεί σε αυτό το σημείο λοιπόν. Το ίδιο και για το άρθρο 28 εξάλλου. Ο κύριος Ροσφόρ είπε ότι είναι ενδιαφέρον. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Όμως έχω αφιβολίες, γιατί και εδώ επικρατεί αβεβαιότητα. Πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο, είτε εδώ, είτε σε μια συνάντηση που θα κάνουμε οι σκιώδεις μεταξύ μας. Κεφάλαιο 5 τώρα. Στο άρθρο 30 αν καταλαβαίνω καλά, περιορίζουμε το εύρο εφαρμογή, το πεδίο εφαρμογή. Το περιορίζουμε σε ορισμένα είδη συμβάσεων. Αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι καλό αυτό ή μήπω πρέπει και τα εξοδομικευμένα συμβόλαια να τα καλύψουμε εδώ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πιστεύω όμως, όπως προτείνει και ο κύριος Χάρμπορ, να έχουμε μία συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών για να μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα νέο κείμενο. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποίησατε αρκετό χρόνο εσεί και καλά κάνατε. Πρέπει όμω και σε εμά να δώσετε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλά. Γι' αυτό και λέω να περιμένουμε μέχρι τι 20 Σεπτεμβρίου. Γιατί έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να το σκεφτούμε καλά και να συνεργαστούμε καλά μεταξύ μα μέχρι τότε. Δεν λέω, υπάρχουν και βελτιώσει. Όμως, πρέπει να υποβάλουμε τροποποίησεις και να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο επόμενο Κιώδης δεν είναι εδώ, αλλά έχω μιλήσει ε, μαζί του και θα σας παρουσιάσω ότι σχόλια θα είχε μαζί με τα δικά μου σχόλια. Λοιπόν, αν κοιτάξουμε το αρχικό κείμενο του κυρίου Σουάπου που είχαμε στην αρχή και είναι κρίμα που δεν το έχουμε μαζί μας σήμερα, αλλά θα το έχετε ίσως εσείς, ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Το σημερινό είναι έτσι πιο μεγαλειώδες. Αλλά δεν, είναι, δεν υπάρχει αντιστοιχεία και αυτό ίσως μας μπερδεύει. Εδώ όταν μιλάτε για πλήρη εναρμόνιση των συγχωνευμένων κεφαλαίων 2 και 3 έχουμε από την άλλη μεριά και τις, ε, την επιλεκτική εναρμόνιση και υπάρχουν και νέες ιδέες στο κεφάλαιο 6 που μας παρουσιάζεται για το πώς η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργάζονται από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια πλήρης εναρμόνιση αλλά μια μεικτή πρόταση. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα χρειαζόμαστε πολύ φαντασία. Σίγουρα το peer review, η αξιολόγηση μεσομοτήμων είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πάντως, όπως λέει η κ. ότι θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιες προϋποθέσεις. Για μένα που είμαι πρόεδρος, βλέπω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν θέλουν προς τα κάτω εναρμόνιση. Δηλαδή, άπαξ και υπάρχει εναρμόνιση, δεν μπορεί αυτή να γίνει προς τα κάτω πουθενά, ώστε να μην πληγεί κανένας καταναλωτής. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι είναι λογικό να προσπαθήσουμε να πετύχουμε εναρμόνιση όπου αυτό είναι δυνατό. Άκουσα τις αναλύσεις σας για τις ρήτρες, της μαύρες και τις γκρίζες όπου καταφέραμε να έχουμε έναν κατάλογο με τέτοιες πρακτικές, τις μαύρες ζήτες και τις γκρίζες. Λέγατε ότι όμως μπορεί να μας μπερδέψει, γιατί για τη μαύρη λίστα μπορεί να συμφωνήσουμε, αλλά μπορεί κάποια πράγματα να υπάρχουν σε μία χώρα στη μαύρη λίστα και σε μια άλλη στην γκριζα λίστα. Και ανάποδα. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο είναι μια προσέγγιση αυτή λογική. Αν όμως έχουμε μια τέτοια προσέγγιση για ρήτρε ε, μαύρης λίστας, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει κάποια αναρμόνιση. ώστε οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα θέτουν σε εφαρμογή τέτοιες διατάξεις στις συμβάσεις τους να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Προτείνω λοιπόν, αν μπορείτε, οι σκιώδεις εισηγητέ με τον εισηγητή μας, να συναντηθείτε από τώρα μέχρι τις 12 Ιουλίου που θα ξαναβάλουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, καλό θα ήταν. 12 Ιουλίου θα προσπαθήσουμε έχοντας το τελικό κείμενο να καταλήξουμε αν μη τι άλλο σε κάποιους στρατηγικούς στόχους. Οπότε μετά θα υπάρχει χρόνος για τροπολογίες. Ελπίζω να συμφωνούν οι σκιώδεις εισηγητές, έτσι θα προχωρήσουμε μόνο. Και η κυρία Γκέπχαρτ τότε θα μπορέσει να ε, στηρίξει την προσέγγισή μας. Και από εκεί και πέρα να μπούμε στις λεπτομέρειες. Αυτό που δεν θα ήθελα, ως πρόεδρος σας το λέω αυτό, είναι να βρεθούμε σε μια θέση όπου υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες ανάμεσα στον εισηγητή μας και τους σκιώδεις εισηγητές όσον αφορά την προσέγγιση. Γιατί πώς θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις λεπτομέρειες. Κύριε δεν με ακούτε, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνετε είναι να συμφωνήσετε για τη δομή της πρότασης. Αυτά τα βασικά στοιχεία που υπάρχουν εδώ και χρησιμοποιώ αυτό το χαρτί, όχι το άλλο, να δείτε πώς θα είναι διαρθρωμένα μεταξύ τους για να προχωρήσουμε σιγά σιγά προς καλά αποτελέσματα. Τροπολογίες θα έχουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αν μη τι άλλο να υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση, ακόμα και αν υπάρχουν διαφωνίες για το επίπεδο αναρμόνισης. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, πιστεύω. Ωραία. Τρία λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Μπορείτε σύντομα να κάνετε τα σχόλιά σας παρακαλώ και αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε μετά την ψηφοφορία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ σύντομα σε ό,τι αφορά τις προτινόμενες τροποποίησεις στα δύο κεφάλαια 4 και 5 ε, θέλω να σημειώσω ότι κατά την άποψη μου υπήρξε πρόοδος προς την απάλληψη της πλήρους εναρμόνισης. Και αυτό έγινε με την εισαγωγή κάποιων διατάξεων που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας εκεί και όπου το κρίνουν σκόπιμο. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να τηρηθεί στην οδηγία και να μην αποτελέσει προϊόν συμβιβασμού αργότερα με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και τώρα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το άρθρο 22, πιστεύω ότι η επιπλέον προσθήκη βάρους για τον καταναλωτή στη διαδικασία επαναχώρησης δεν είναι προς το συμφέρον ούτε των καταναλωτών ούτε των εμπόρων ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει άμεσα το δικαίωμα της αποζημίωσης αν ο έμπορος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ο καταναλωτής θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια δικαίου κατά τις συναλλαγές του. Στο άρθρο 26 πιστεύω ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν στις παραγράφους 1 και 2 είναι ορθές και προσθέτουν σαφήνεια στο κείμενο. Όμως η παράγραφος 5α η οποία περιορίζει τη δυνατότητα του καταναλωτή να επαναχωρεί στις περιπτώσεις μικροβλαβών αποτελεί προβληματικό σημείο. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιο καθορίζει το τι αποτελεί μικροζημιά. Με βάση ποια κριτήρια θα προσμετράτε το μέγεθος της ζημιάς. Ε, στο άρθρο 28 είναι πολύ σημαντική η προσθήκη της δυνατότητας των κρατών μελών να επεκτείνουν τη διάρκεια εγγύσεων πέραν των δύο ετών. Θα πρέπει όμως να ξαναδούμε τη διαγραφή που προτείνεται από τον εισηγητή για την ανανέωση της περίοδου εγγύησης όταν υπάρξει αντικατάσταση του προϊόντος. Και τέλος, σχετικά με το κεφάλαιο 5, η ελάχιστη εναρμόνιση είναι ορθότερη από το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Η μόνη προσθήκη που θα πρέπει να μελετηθεί είναι η ισχυροποίηση των ρητρών που θεωρούνται καταχρηστικές σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ο μαύρος κατάλογος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Okay. Uh, thank you very much indeed. Um... πολύ. Από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η κυρία Βόλης τώρα θα μας πει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση για να παραστώ σήμερα και να μιλήσω για αυτό το θέμα. Είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Σβάμπ για τη σκληρή δουλειά του. Για τη δική μας Επιτροπή τώρα θεωρούμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά τη συνολική εικόνα, ούτως ώστε όλες οι ψηφίδες να κολλάνε εκεί που πρέπει. κάποια προκαταρτικά σχόλια μετά τη σημερινή συζήτηση. Αν θέλουμε να φτάσουμε ε, εκεί που πρέπει να φτάσουμε, ε, πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ. Τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα και συμφωνώ ε, με σας, Πρόεδρε, ότι αν δεν συμφωνήσουμε για τη δομή, θα είναι αδύνατο το έργο μας να προχωρήσουμε και να βρούμε μία λύση. Τώρα, για τη δική μας ε, Επιτροπή, θέλω να σας πω τα εξής. Σε λίγο ε, θα παραστούμε στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων ε, για, τις, για το δίκαιο των συμβάσεων. Οι, οι εμπειρογνώμονες λένε ότι πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών συνολικά σε όλες τις συμβάσεις. Αλλιώς δεν θα επιλεγεί αυτό το εργαλείο ως προαιρετικό εργαλείο. Θα ήθελα να κάνω μια τελική υπόδειξη. Διάφοροι ομιλητές ανέφεραν το βρετανικό δικαίωμα απόρριψης. Και ορισμένοι θεώρησαν ότι υπάρχει παναχώρηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αναφέρθηκαν και άλλα παραδείγματα, ένα γαλλικό παράδειγμα κτλ. Θα πρέπει να δούμε πού υπάρχει παναχώρηση ή πού κολλάμε. Ε, να έχουμε ένα κατάλογο με, όλα τα, με όλες τις υπαναχωρήσεις, ε, να δούμε αυτά τα δύσκολα θέματα για να προσπαθήσουμε από εκεί να σημειώσουμε πρόοδο. Μπορεί να είναι μακρύ αυτό ο κατάλογο, αλλά θα πρέπει να τον, να τον επιλύσουμε, να βρούμε λύση για όλα αυτά τα σημεία που είναι δύσκολα, που κολλάμε. Ευχαριστώ την ε, κυρία Γουόλη. Ε, τον έχουμε αυτόν τον κατάλογο. Από, την, ε, από προηγούμενο, ε, προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Γιατί ζητήσαμε από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ε, να μας τον δώσει. Επίσης, για το κοινό πλαίσιο, αυτό που είπατε, το άκουσα. Νομίζω υπάρχει και στη δομή που μας παρουσίασε ο Ανδρέας Βάμπ. Ο εισηγητής δεν με ακούει. Ανδρέας, μπορείς να με ακούσεις. Μιλούσα για αυτή την αναφορά στο κοινό πλαίσιο που την έχει εντάξει στη δομή που μας παρουσίασε. και ίσως θα πρέπει μια ενδιάμεση α, διευθέτηση για να υπάρξει αυτό το πλαίσιο να μπει στο κεφάλαιο 6. Πριν περάμε στην ψηφοφορία για τις δύο εκθέσεις, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σημαντικό ε, σημείο που συζητήσαμε στη συνεδρία των συντονιστών. Παρακαλώ να ησυχάσετε. Παρακαλώ, ησυχία. Με βάση τη ε, διαδικασία της επιτροπολογίας, είμαστε υπεύθυνοι ως Επιτροπή για όλες τις προτάσεις ε, για τα εφαρμοστικά μέτρα που εκπονήσαμε εμείς και το προηγούμενο Κοινοβούλιο. Ε, είπαμε με βάση τη διαδικασία να κοιτάξουμε τα εφαρμοστικά μέτρα στη συνεδρία των συντονιστών. Ε, θεωρούμε μερικές φορές ότι έχει υπερβολικές εφαρμοστικές ε, αρμοδιότητες και το μέτρο δεν είναι συμβατό με το στόχο ή το περιεχόμενο του βασικού εργαλείου, αρχική νομοθεσία, ή δεν σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Ο εφαρμοστικός κανονισμός λοιπόν για τα προϊόντα φώκιας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πέρασε από το ε, περασμένο κοινοβούλιο υπό την ηγεσία της κυρίας Βόλης που ήταν συγγήτρια. Η Κομισιόν μας έστειλε ένα σχέδιο εφαρμοστικών μέτρων. Στις 19 Μαΐου το λάβαμε και μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουμε, την έχουμε αυτή την προθεσμία για να το κοιτάξουμε. Όμως ο ίδιος ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 2010. Σε δύο μήνες δηλαδή. Επομένως, θα πρέπει να εγκρίνουμε νωρίτερα τα εφαρμοστικά μέτρα, ούτως ή άλλως. Το συζητήσαμε χθες με την Κομισιόν στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών και οι συντονιστές εξέτασαν την θέση ε, και ψήφισαν με μία αποχή να συστήσουν ότι δεν αντιτιθέμεθα στα εφαρμοστικά μέτρα και θέλουμε να, το, να εγκριθούν αυτά το συντομότερο δυνατόν, το νωρίτερο δυνατόν, ούτω ώστε όταν τα πλήρη μέτρα στις 20 Αυγούστου τεθούν σε ενισχύ για τα προϊόντα φώκιας, τότε και τα εφαρμοστικά μέτρα θα είναι σε, θα είναι σε λειτουργία και θα τα συνοδεύουν. Θέλω λοιπόν σε λίγο να ψηφίσουμε τα σχετικά μέτρα, αλλά θέλω να πω στην κυρία Γουόλης που ήταν η συγγήτρια ε, να μας μιλήσει γιατί γνωρίζει πολύ καλύτερα τον κανονισμό οποιονδήποτε άλλο. Κανονισμός για τα προϊόντα αυτο, ε, φώκιας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξοικειωθήκαμε με το θέμα. Την περασμένη Δευτέρα συζητήθηκε διαμακρών από όλες τις ομάδες για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο. Είναι περίπλοκο, χρειάζεται πολύ προσεκτική εφαρμογή για να βεβαιωθούμε ότι κάποιοι θα μπορούν να προστατεύουν τις κοινότητές τους και τη δυνατότητα να συνεχίζουν τις ε, διαδικασίες αυτές. Ε, το... Οι εμπορικές δραστηριότητες ε, έχουν περιοριστεί τώρα, έχουν σταματήσει. Έτσι λοιπόν οι εκτελεστικοί εφαρμοστικοί κανόνες έπρεπε να σχεδιαστούν προσεκτικά και ακούσαμε λεπτομερώς από την Κομισιόν τι έκανε για αυτό το θέμα και από πού άντλησε ιδέες, από ποια παρόμοια νομοθετήματα. Η λεπτομερής έκθεση επίσης πρόκειται ανεξάρτητα να κρίνει να αξιολογήσει τους εφαρμοστικούς κανόνες. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι έκαναν πολύ ισορροπημένη και προσεκτική δουλειά. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, νομίζω, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπατε, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μην σκεφτεί να απορρίψει τους εφαρμοστικούς κανόνες, γιατί κάτι τέτοιο θα μας έβαζε σε πολύ δύσκολη θέση. Επίσης, η ημερομηνία θέση σε ισχύ που ήθελε η Κομισιόν είναι ο Αύγουστος, πολύ κοντά. Οπότε αν κάναμε κάτι τέτοιο θα παρεκκλίναμε από την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Επίσης πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και λόμπιστς ζητούν να τεθεί σε ισχύ αυτό το νομοθέτημα και του χρόνου, το 2011, θα μας υποβάλει έκθεση κομισιών, οπότε το, έχουμε προστασία. Και το καλύτερο είναι να το βάλουμε να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, οπότε εγώ συνιστώ θετική ψήφο στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτ ε, είπε ότι θέλει να μιλήσει, παρόλο που δεν είχα προβλέψει μακρά συζήτηση για το θέμα. Ορίστε. Ευχαριστώ. στην ομάδα μου συστήνω να απόσχει και πρέπει να το δικαιολογήσω για να ξέρει ο κόσμος περί πρόκειται. Χθε το βράδυ και στη συνεδρίαση των συντονιστών απέσχων γιατί η διαδικασία αυτή δεν μου φάνηκε αρκετά σαφής. Δεν καταλαβαίνω γιατί στους εφαρμοστικούς κανονισμούς το κείμενο του κανονισμού μάλλον, όχι της οδηγίας, λαμβάνεται ε, σε διαφοροποιημένη μορφή και κάποιοι τομείς έχουν μείνει απ' έξω. Δεν κατάλαβα τη διαδικασία. Δεν ψήφισα κατά γιατί σε μια ερώτηση του Προέδρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε καθαρά. Η ερώτηση ήταν του Πρόεδρου ενώ στο αρχικό κείμενο του κανονισμού στο άρθρο 3 υπάρχει ξαφής ε, διατύπωση που ισχύει ως βάση για τους εφαρμοστικούς κανονισμούς και η Κομισιόν είπε ναι οπωσδήποτε και γι' αυτό είπα και εγώ εντάξει δεν θα απορρίψουμε αυτούς τους ε, εφαρμοστικούς κανόνες, αλλά μου παραμένει μια βεβαιότητα Γιατί στους εφαρμοστικούς κανόνες επιλέγεται διαφορετική διατύπωση από την οδηγία καθ' αυτή. Γιατί το κάνουν αυτό. Και γι' αυτό συνέστησα στην ομάδα μου την αποχή. Ε, ε, δεν, ήθελα να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση, συνάδελφοι, αλλά εάν υπάρχει ενδιαφέρον και θέλετε συζήτηση, θα πρέπει να γίνει σήμερα το απόγευμα, γιατί το πρωί θα πρέπει να ψηφίσουμε. Η κυρία Ρούλερ, η κυρία Ρόιτερ, φαντάζομαι και άλλοι θα ζητήσουν το λόγο. Οι συντονιστές το έχουν συζητήσει και φαντάζομαι ότι θα έχουν, έχουν καταλήξει συστάσεις. Ξέρω ότι ήρθαν οι κανόνες καθυστερημένα, αλλά όπως είπε και η κυρία Βόλς είναι σημαντικό να το συζητήσουμε σήμερα. Οπότε η Γραμματεία θα διαθέσει όλα τα έγγραφα και μετά θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα στις 4.30 το θέμα σε πλήρη σύνθεση της Επιτροπής, γιατί άλλη ευκαιρία δεν έχουμε για να μπούμε στις λεπτομέρειες, εκτός και αν θέλετε να προχωρήσω στην ψηφοφορία χωρίς άλλη συζήτηση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θέλετε και άλλη συζήτηση. Οπότε θα προσθέσουμε σήμερα το απόγευμα ένα ακόμα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν λεπτομέρειες των εφαρμοστικών κανόνων στο website όπως και όλο το κείμενο. Μπορεί να μιλήσουν κι άλλοι και αμέσως μετά θα ψηφίσουμε. Οπότε, εάν θέλετε να ψηφίσετε, θα πρέπει να έρθετε στις 4.30 το απόγευμα. Συμφωνούν όλοι. Εντάξει. Αποφασίσαμε λοιπόν και η κυρία Βόλης. Τι ώρα θα, είναι, ε, θα γίνει η ψηφοφορία. Εξαρτάται από το πόσο θα πάρει η συζήτηση. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά αν θέλετε να ψηφίσετε πρέπει να έρθετε στη συζήτηση που θα αρχίσει στις 4.30. Συγγνώμη, αλλά είναι δυνατόν να έρθει και η Κομισιόν και να εξηγήσουν αυτά που εξήγησαν και χτες το βράδυ. Προφανώς θα προσκαλέσουμε την Κομισιόν και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να έρθει. Ο κύριος Ροσφόρ, προτείνω να ψηφίσουμε τώρα. Let's, let's find Για να δούμε. Υποστηρίζετε από την πλειοψηφία η πρότασή σας και τότε. Εντάξει, κυρία Ρούλερ, να πω κάτι. Δεν είναι καλό το πώς μεθοδεύονται τα πράγματα. Κύριε Χάρμπορ, ξέρετε ότι η συγγήτρια τότε ήταν στη μειοψηφία, στην ψηφοφορία και η άποψή της δεν καλύφθηκε από την Επιτροπή. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι οι συγγητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και ίσως ε, μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο μιλία για όλους. Δεν μπορεί όμως να μιλήσει η συγγήτρια μόνη εκ μέρους της Επιτροπής, συγγνώμη, αλλά η διαδικασία δεν είναι σωστή. Καλά. Δεν μίλησε η συγγήτρια, τη γνώμη της ζήτησα γιατί ήταν ε, η συγγήτρια. Η Επιτροπή θα ακολουθήσει ή θα αποφασίσει. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε. Τι θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε αν θα ψηφίσουμε τώρα. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι καλύφθηκαν από τη συζήτηση ή έκαναν τις παρεμβάσεις τους. Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι το καλύτερο να το κάνουμε το απόγευμα. Ο κύριος Σβάμπ. Ναι, αλλά το μεσημέρι δεν θα είναι όλοι. Δεν θα έχουμε απαρτία. Ίσως τον Ιούλιο, ίσως έρθουν μερικοί, αλλά είναι δύσκολο για μας. Το πρόβλημα με την αναβολή είναι ότι δεν θα έχουμε χρόνο πια. Αυτή είναι η δυσκολία. Δεν μπορούμε να πάμε Ιούλιο εύκολα. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που είχαμε να το συζητήσουμε. Ε, γι' αυτό λέω το απόγευμα, γι' αυτό το έβαλα και σήμερα μετά τις χθεσινές συζητήσεις των συντονιστών. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει εναλλακτική. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Λοιπόν, έτσι μου φαίνεται ότι θα το πάμε για 4.30 σήμερα το απόγευμα. Φωνάξουμε και την Κομισιόν και θα ε, ελπίζω να είστε και όλοι εσείς ε, εκεί τότε για να ψηφίσετε. Κύριε Σαρίας. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αλλάξω τα σχέδιά μου. Εγώ φεύγω, πάω στην Ισπανία σήμερα το απόγευμα. Οπότε αν θέλετε να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, τουλάχιστον να μην ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα, να ψηφίσουμε κάποια άλλη στιγμή για να είμαστε όλοι παρόντε. Πρόεδρο. δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Τέλο πάντων, Κρίστα Μπουζόη. Πρόεδρε, πρότεινα να ψηφίσουμε τώρα. Μπορείτε να το θέσετε σε ψηφοφορία για να δούμε αν υπάρχει πλειοψηφία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, αν η πλειοψηφία θέλει να ψηφίσουμε τώρα, να ψηφίσουμε τώρα. Αν όλοι οι συντονιστές είχαμε μιλήσει και αν σε μισό ή ένα λεπτό κάθε ομάδα είχε πει τη γνώμη της, θα είχαμε τώρα προπολού αρχίσει την ψηφοφορία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το, τα κάνουμε αυτά. Θα δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση. Λοιπόν, οι συντονιστές. Ωραία, κυρία Κέπαρτη, κυρία Ρούλε, <clears throat> να μας εξηγήσουν τις θέσεις τους. Η κυρία Ρούλε πρώτα. Συντομότατα, λέω να ψηφίσουμε υπέρ στην ομάδα μου, γιατί υπάρχουν και ο κίνδυνος οι κανόνες να ε, ε, μην εφαρμόζονται. Η Κομισιόν μας εξήγησε δύο σημεία που με έπεισαν άλλωστε. Το ένα σημείο και γι' αυτό είπα να ψηφίσει η ομάδα μου υπέρ. Το ένα είναι ότι το νομικό κείμενο παραμένει η νομική βάση, το αρχικό που είχαμε ψηφίσει και το δεύτερο ότι στις 12 Αυγούστου επιτέλους θα αρχίσει να εφαρμόζεται γιατί αλλιώς το φθινόπωρο θα είμαστε στην, στην ίδια δυσκολία, αρχίζει το κυνήγι στο Καναδά και θα ε, μας παραπονούνταν ότι δεν κάναμε τίποτα. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή να ψηφίσουμε, να κλείσει το θέμα και το 2011 έτσι κι αλλιώς θα μας υποβληθεί και η έκθεση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κύριε Σουάμπα, όχι. Επίτε μας τη θέση σας. Συμφωνώ απόλυτα με την θέση της κυρίας Ρούλε. Ρούλε. Είχαμε χθες μια συζήτηση και ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητο το θέμα. Ξέρω ότι μας έστειλαν email, διάφορες ε, φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αλλά τώρα η ιδέα δεν είναι να ξαναρχίσω με τη συζήτηση για τις ε, φώκες και το ε, εμπόριο και αν επιτρέπεται ή όχι, γιατί αυτό το αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε αν ο αρχικός κανονισμός εφαρμόζεται καλά με τον καινούριο και αν έχουμε και η μικρή Κινταϊάννα Ουόλης χθε εξήγησε τις διαδικασίες, χρειάζεται πολύ έγκυρος λόγος για να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν. Και ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι θα τεθεί ο κανονισμός σε εφαρμογή τον Αύγουστο, οπότε δεν λύνουμε πολλά αν αντιταχθούμε τώρα. Γι' αυτό λέω να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία και να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, τώρα μίλησαν όλοι οι συντονιστές που ήταν χθες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ας ψηφίσουμε. Συμφωνούμε με τη σύσταση των συντονιστών να μην ταχθούμε κατά των εφαρμοστικών μέτρων. Περ, κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο η Επιτροπή συμφωνεί ότι πρέπει να ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να το εγκρίνουν τον Ιούλιο πριν ε, τεθεί σε εφαρμογή το, η οδηγία. Υπέρ, κατά, δεκτό και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν κάποιος θέλει λεπτομέρειες, υπάρχουν και αυτές. Προχωρούμε. Είπαμε για ηλεκτρονική ψηφοφορία, επειδή έχουμε πολλές, οπότε για να ελέγξουμε λίγο τα νούμερα καταρχήν, αν έχετε όλοι τις κάρτες σας. Για το ΕΛΚ πρώτα απ' όλα ποιοι ψηφίζουν. Μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη του ΕΛΚ παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες πόσους έχουμε. 12. 14 θα πρέπει. Ξανά, άλλη μια φορά. Για το ΕΛΚ. Ψηφίστε. Ωραία, 14 έχουμε τώρα. Α, 15 έχουμε τώρα. Όποιος ήταν ο τελευταίος. Ένας δεν πρέπει να ψηφίζει. Ο κύριος Καράς δεν θα ψηφίζει, εντάξει. Άλλοι από το ΕΛΚ που θέλουν να ψηφίσουν και δεν μπορούν, να το ξέρουν, ε. Εσείς χει, καλά. Ποιοι είναι υπέρ από το ΕΛΚ, είμαστε εντάξει, είμαστε εντάξει. Όχι, ξανά, η ΕΛΚ. Υπέρ. Τώρα. Για να ελέγξουμε. Τελικός έλεγχος. Πάλι 15. Ένας από εσά δεν πρέπει να ψηφίζει. 14 έχουμε τώρα, εντάξει. Για τους σοσιαλιστές τώρα. Υπέρ, σοσιαλιστές. Ψηφίστε παρακαλώ. 8. Θέλετε ενισχύσει. Ωραία, για του υπόλοιπου φαντάζομαι είναι εντάξει. Τέσσερι φιλελεύθερου κλπ. κλπ. Εντάξει, λέει ο πρόεδρο, ξεκινάμε. Έκθεση του κυρίου Τρασκόφσκι για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Τσασκόφσκι μήπως πριν ξεκινήσουμε. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν. Τίποτα άλλο. Παράγραφος 7. Ψηφίζουμε. Προπολογία, αριθμός 1 του κύριο Κρότσμαν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμό 2 Το κ. Κρότσμαν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Έχουμε προφορική τροποποίηση. Υπέρ παρακαλώ. Είναι στους φακέλους σας. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10α Τροπολογία αριθμός 3 του κ. Τρασκόφσκη και του κ. Καρά με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά εγκρίνεται. Κατά πίπτη 3. 10α νέα με προφορική πάλι τροποποίηση υπέρ κατά εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 12α. Τροπολογία 5 με προφορική τροποποίηση Τρασκόφσκι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 πίπτη. 6 τώρα. Κρότσμαν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 Κρότσμαν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 με προφορική τροποποίηση του κ. Κρότσμαν υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 Κρότσμαν υπέρ κατά εγκρίνεται. 10 με προφορική τροποποίηση του κ. Τρασκόφσκι υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 10 καταπίπτει. Τροπολογία 11 του κ. Τρασκόφσκι υπέρ κατά εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 32 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Τρασκόφσκι. Τώρα περνάμε στην έκθεση του κυρίου Άριας. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο εισηγητή θέλει μήπω να πει κάτι πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους κατά τη σύνταξη του σχεδίου αυτού έκθεσης και για όλου του συμβασμού του οποίου μπορέσαμε και καταλήξαμε για αυτή την ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και όλα τα μέλη της Γραμματείας εδώ της Επιτροπής μας και τις πολιτικές ομάδες, τους βοηθούς τους κλπ. Ωραία, ψηφίζουμε λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 49, υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται. 50 και 56 είναι ίδιες, υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 51, Λουιγκρές, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 Κέλλη, παράγραφος 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολίγιο 53 Μακλάρκιν. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 54 Κονέλης Δεγιόν. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 59 διάφοροι συνάδελφοι, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 55 τώρα, Λόκεγκαρτ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 58. De Jong. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57. Κορέα Δεκάμπος υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μια συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Που σημαίνει ότι πάμε μετά την 61, 60 και 62 που καλύπτονται συμβαστική, στην και 64, ναι. Πάμε στην... 66. Ροσφόρ. Διαμαρτυρίες από την αίθουσα. 62. Δεν ήταν συμβαστική, όντω. 62. Ποιοι είναι υπέρ τη 62, παρακαλώ, του κ. Ντεγιόν. Κατά. Απορρίπτεται. 66. Α, 65. Ε, δεν τα έχω καλά τότε. 65 λέει ο πρόεδρος. Ωραία, συγγνώμη. 65. Τούρνεν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 66 του κυρίου Ροσφόρ. Αλλά κατά τμήματα ψηφοφορία είναι αυτή. Πρώτο τμήμα. Τη τροπολογίας 66 υπέρ Α, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 66. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τις τροπολογίες 66 τώρα. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της 66. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22-12. Τώρα, τροπολογία 68. Σβάβου. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 68. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 67. 69 is next. Uh, so, 69 uh, υπέρ, uh, uh, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία Ήτρε τώρα, παράγραφος 13 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάντα Ήτρε 30 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 6 τώρα, τροπολογία 70. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 71. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Νομικής Επιτροπής, παράγραφος 11. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, Νομικής Επιτροπής υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογίες 72 και 73 που είναι ίδιες υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Κυρία Σκόβολα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 75. Είναι γλωσσική, οπότε δεν την ψηφίζουμε. Νομική επιτροπή τώρα παράγραφο 1. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 77 του κ. Κορέντε Κάμπος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 78 του συγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Νομικών υποθέσεων, παράγραφος 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 15 Παντανομικής Επιτροπής υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 3 της Ήτρε υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στη συμβαστική τροπολογία αριθμός 2. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά, εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην Ήτρε, παράγραφος 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα την 13 της Γιούρη ως προστίκη υπέρ, κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 8α 8α9. Τροπολογίες 84, 85 και 98 που είναι υπέρ, κατά εγκρίνονται. Ήτρε 15 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τροπολογία 86 υπέρ που είναι προστίκη. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 86 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορίας εγκρίθηκε 21 ψήφι υπέρ, 13 κατά. Ήτρε 31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 90, έχει αποσυρθεί. 91 τώρα, τέρνου είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 92, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμό 4 υπέρ παρακαλώ. Κατά εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία... Νομικών υποθέσεων 16 και 4 προς υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά θα ελέγξουμε. Τροπολογία 101. Λοιπόν, ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 22 υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 102. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. 18 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 99 του κ. Ντεγιόν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 100 του κ. Κρότσμαν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 103 του κ. Γκρέκ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική τροπολογία αριθμός 5 στην 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οπότε πάμε τώρα στην τροπολογία αριθμός 110 του κ. Ντεγιόν ως προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Κέλλη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 114 Κέλλη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα τις τροπολογίες της Ήτρενα, να τις μαζί. 16, 18, 19, 20 και 21 μαζί. Υπέρ. Όχι. Δεν θέλετε. Ναι. Ωραία. Όλες μαζί. On block λοιπόν. 16 με 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 116. Στην παράγραφο 12 υπέρ. Α, όχι. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 116. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη προφορίες, Εγκρίθηκε 20 υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 115 Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε. Παράγραφος 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 120 τώρα. έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 118. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Θα ελέγξουμε. Τροπολογία 117. Μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 12 κατά. Τροπολογία 119 είναι γλωσσική τροπολογία. Δεν την ψηφίσουμε. Παράγραφος 16α ναι. 121, 124, 122, 123 υπέρ παρακαλώ. Κατά εγκρίνονται. Νομικών υποθέσεων. Παράγραφος 14 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ήτρε, αριθμός 1 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 125 τύρινεν υπέρ, κατά, νομικών υποθέσεων 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Νομικών υποθέσεων 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 126 τύρινεν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα των νομικών υποθέσεων την 5, την 6 και την 10 μαζί να τις ψηφίσουμε, εντάξει. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Όχι. Α, δεν θέλετε μαζί. Αν μπλοκ. Τι είπατε. Όχι μπλοκ. Καλά. No block. Χωριστά. 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127 της κυρίας Τούρινεν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 128 του κυρίου Ροσφόρ και Κρόσμεν. Υπέρ. Να ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ για την 128 Ροσφόρ. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, 21 ψηφί κατά. Τροπολογία 129, Ζουβάν και Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 129. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 16 κατά. Ήτρε τώρα, παράγραφος 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 130, 131 και 132 υπέρ παρακαλώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ 130, 131 και 132. τη ψηφοφορία. Εγκρίνονται 26 υπέρ 7 κατά. Τροπολογία 133 έχει αποσυρθεί. 134 τώρα. Κρότσμαν και Μάντερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομικών υποθέσεων 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 136 Κρότσμαν. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 136 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνονται 20 υπέρ 13 κατά. Τώρα 135 και 137 μαζί ως προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνονται. Ε, 5 υπέρ, ήτρε δηλαδή, υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 139. Κρέκ. Ξεκινάει ψηφοφορία 139 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Κατά. 138 Τύρνεν. Ξεκινάει ψηφοφορία ηλεκτρονικά πάλι για την 138. Ψηφίστε. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19 κατά. 15 υπέρ. Νομικών υποθέσεων παράγραφος 19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομικών υποθέσεων 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 142 που δεν περιλαμβάνεται στον συμβιβασμό. Υπέρ παρακαλώ της 142 κατά απορρίπτεται. Τώρα νομικών υποθέσεων 18 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 146 υπέρ κατά εγκρίνεται. 148 του συγκητή υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα μπορούμε τις επόμενες να τις δούμε μαζί, νομικών υποθέσεων και ήτρε. Ωραία. Είναι ήτρε 9, 23, 26, 29 υπέρ κατά εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 7 τώρα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην Ήτρε, παράγραφος 12. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομικών υποθέσεων 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 153 τώρα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και ερχόμαστε τώρα στη συμβαστική τροπολογία αριθμός 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα. Παράγραφο 8. Ήτρε. 8, 10, 24, 28. Όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 158 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 160. Αυτή καταπίπτει. 159. Ηλεκτρονική ψηφοφορία να κάνουμε καλύτερα για αυτήν. «159 υπέρ, κατά». Σαφώς περνάει. Ήτρε, παράγραφος 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 161. De Jong. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 164-165 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 166-163 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 162. Αρχές ψηφοφορίας παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 19 κατά. Πάμε στα εκτιμώντας τώρα, σε θεωρητικές σκέψεις. Τροπολογία 14, στο υπέρ κατά εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. 16 και 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 20 και 21 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Γιούρι, εκτιμώντας α υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήτρε, εκτιμώντας α υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας γ 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήτρε, ε, εκτιμώντας β υπέρ, κατά εγκρίνεται. Πάμε τώρα. Για το ΔΕΛΤΑ και το Ε μαζί. Για τα το ΔΕΛΤΑ και Ε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα. 23. Τροπολογία 23. Κορέα Ντεκάμπος υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 και 25. Αυτές καταπίπτουν. Πάμε στην ίτρε C. Γ. Δηλαδή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά εγκρίνεται Γιούρι εκτιμώντας β υπέρ κατά εγκρίνεται Ήτρε εκτιμώντας J υπέρ κατά εγκρίνεται ε νέο τροπολογία 8, 28 υπέρ κατά εγκρίνεται 30 υπέρ κατά εγκρίνεται. 29 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα τις υπόλοιπες on block, υπέρ κατά εγκρίνονται αυτές τις επο, επόμενες τρεις DJ και F. Τροπολογία 31 υπέρ κατά εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, Γιούρι ε, ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 39 υπέρ. Ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Για 39. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, 14 κατά, 41. Τροπολογία 41. Υπέρ. Ε, ξεκινάμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 41. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 κατά, 14 υπέρ. 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 19 κατά. 38. 38. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένα ψηφοφορία. Πέρας. Καταπίπτει επίση. 16 υπέρ, 18 κατά. Τώρα, έχουμε μαζί τις Γιούρι F, G, I και J υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 43 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε, H, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 45, Κρότσμαν υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 46, Μακλάρκιν, με ψηφορή κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, Τη 46 υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Τη 46. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα έναξη ψηφοφορία. Πέρα. Α, είστε πολύ αργοί. Πέρα ψηφοφορία τώρα. Εγκρίνεται 22 υπέρ, 7 κατά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα της C H και της ε, I μαζί, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 47 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 48 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Πάμε στις αναφορές. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Πάμε στο σχέδιο έκθεσης συνολικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία συνολικά για την έκθεση. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 32 υπέρ και καμία ψήφος κατά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ρίας ε, Σεβερή, ευχαριστώ τους κοιόδης συγγητές. Ε, Νομίζω ότι θα είναι σημαντική η έκθεση αυτή για τη δουλειά μας. Όσοι θέλουν να φύγουν μετά το τέλος της να φύγουν ήσυχα. Τώρα έχουμε ένα δίλημα. Έχω 8 ε, ομιλητέ, ε, συν την Κομισιόν που θέλουν να μιλήσω για την έκθεση ΣΒΑΜΠ. Και επίση θέλω να επιτρέψω στον κύριο Σαντεμόζε να ξεκινήσει τη δική τη ε, έκθεση και έχουμε και τη συνεδρίαση των συντονιστών σε 10.30. Κύριε Σανταλμόζε, δεν μπορείτε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Ιουλίου, σωστό? Σωστό γνέφει, κυρία Σκαλτεμόζε. I mean, I would rather give you more time. Alternatively, if you want to launch... Αν θέλετε σύντομα να μιλήσετε για την έκθεσή σας, μπορείτε. Uh, well, can I propose the following? Um, I think... Προτείνω το εξή. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να κάνουμε και πλήρη συζήτηση με τους σκιώδει ηγητέ, αλλά ξέρω ότι θέλετε να μας πείτε αρχικά έτσι, τις σα σας ιδέες τουλάχιστον. Λοιπόν, έχουμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Είτε θα αφήσουμε την έκθεση ΣΒΑΠ για τις 12 Ιουλίου ή θα δώσω σε όλους ένα λεπτό για να μου μιλήσουν, να μου πούν τι θέλουν για την έκθεση ΣΒΑΠ και να έχουμε λιγότερο χρόνο για την έκθεση ε, Σκαλντεμόζε. Κύριε Σβάμπ, με ακούτε, να σας πω τι θα κάνουμε. Γι' αυτό σας το λέω δηλαδή. Λοιπόν, θα δώσω σε κάθε ένα από τους κάτω... Ο κύριος Αρίας έφυγε, ο κύριος Λάγκ είναι εδώ. Όλοι αυτοί θα μιλήσουν από ένα λεπτό. Έτσι για να σχολιάσουν την έκθεση ΣΒΑΠ και μετά θα δώσω την, το λόγο στον κύριο Πράγκ. Λίγο μετά τις 11 θα πρέπει να έχουμε κλείσει ε, την έκθεση ΣΒΑΠ και μετά θα έχουμε μισή ώρα για την έκθεση Σκαλντεμόζε. Και κύριε Σουάπ, και εσείς, πολύ λίγο στο χρόνο, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τον εισηγητή. Μιλάμε για τη δομή και την προσέγγιση. Ε, ακούσαμε μόνο η τοπάθεια, ότι όλα επιδεινώνονται, είναι απαράδεκτα. Και ποια είναι η άποψη δηλαδή, των σοσιαλδημοκρατών, ποια είναι η πρότασή του, ποια είναι η φιλοσοφία του. Γιατί ακούσαμε ε, συγκριτική ανάλυση με το γαλλικό δίκαιο και με το γερμανικό δίκαιο, αλλά είμαστε 27 κράτη-μέλη, σα ε, υπενθυμίζω. Δεν είναι μια νομική εδώ πέρα προσπάθεια για να συγκρίνουμε τις νομοθεσίες. Προσπαθούμε να έχουμε ένα γενικό όραμα, καλύτερη προστασία για τους καταναλωτές και τελικά να κερδίσουν όλοι, και οι καταναλωτές και οι, μικρότερες, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Γκέπχαρτ, και πού είναι το όραμά σας δηλαδή εσάς? Δεν είναι εισηγήτρια κυρία Γκέπχαρτ, λέει ο πρόεδρος. Δεν θα της επιτρέψω λοιπόν να απαντήσει. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Ο κύριος Λέχνα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να πω και εγώ κάτι. Κατανοώ αυτά που είπε η κυρία Γκέμπχαρτ, αλλά κυρία Γκέμπχαρτ παραβλέπετε ότι η εναρμόνιση είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή και εσείς είστε ευρωπαίστρια. Ας... Τώρα αν είναι βισκασέ ή δικαίωμα επαναχώρησης αυτά δεν θα αν δεν τα πειράζουμε αυτά καθόλου, τότε ας παρατηθούμε από την προσπάθεια. Δεν ξέρω, εγώ έχω κάθε σεβασμό στα γαλλικά βίσκασε, όχι επειδή τα θεωρώ σωστά, επειδή σέβομαι τις εθνικές παραδόσεις, ε, παραδόσεις στο δίκαιο, στους πολίτες. Αλλά επειδή είναι σύνθετο το αντικείμενό μας, πιστεύω ότι η πρόταση βελτιώνει λίγο τα πράγματα. Η οδηγία για τα καταναλωτικά αγαθά έχουν σχέση βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει με την καταχρηστική ρήτρα της σχετικής οδηγίας. Ε, μπορούμε να τα δούμε και διαφορετικά, να τις δούμε χωριστά. Αλλά έτσι θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο Παρακολουθώ τη συζήτηση και βλέπω ότι γυρίζουμε σε κύκλους και επαναλαμβανόμαστε. Αν δεν συμφωνούμε, τότε να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό που ίσχυε πριν και όχι στην πρόταση της Κομισιόν και να προχωρήσουμε πιο σιγά, σταδιακά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ περίπλοκη αυτή η προσπάθεια. Και αντί για κάτι τόσο περίπλοκο, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε μια σωστή ισορροπία από τη μία να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε βεβαίως αυτά τα δικαιώματα να τα χρησιμοποιήσουμε για να υποσκάψουμε τα... το σθένος ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να ενδυναμώσουμε και την ενιαία αγορά. Πρέπει να δουλέψουμε με τέτοιον τρόπο ότι τα οικονομικά του συμφέροντα προστατεύονται. Μιλάμε για την ενοποίηση των ε, κλασικών δικαιωμάτων. Ο κ. Ζουβά. Πρόεδρε, ξέρω ότι δεν είσαστε μάγος, αλλά το κείμενο μας ήρθε πολύ καθυστερημένα, είναι περίπλοκο και μας δίνεται και ένα λεφτό να μιλήσουμε. Τι ανταλλαγή απόψεων αυτή. Θεωρητικά ανταλλάσσουμε απόψεις. Τέλος πάντων, τούτου λεχθέντος. Το κείμενο είναι περίπλοκο και στις επικρίσεις μας για τη δουλειά των, του εισηγητή να δείξουμε ταπεινοφροσύνη. Γιατί εγώ με ένα τέτοιο κείμενο δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω ως εισηγητής. Ιδανικά θα έπρεπε τα συστήματα να είναι εναρμονισμένα πλήρως. Οι, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να έχουν ένα κανόνα να σεβαστούν. Αλλά δεν υπάρχουν ιδανικέ ε, συνθήκε, γι' αυτό πρέπει να μπαλώσουμε από εδώ και από εκεί. Γιατί δεν υπάρχουν ιδανικέ συνθήκε, έχουμε διαφορετικέ παραδόσεις κτλ. Και ο εισηγητή είναι εδώ για να βρει τη λιγότερο κακή λύση και πρέπει να το τιμήσουμε αυτό που κάνει, αυτό το έργο του. Ε, αυτό το σχέδιο είναι προστασία, ονομάζεται προστασία του καταναλωτή. Επομένω, το τελικό κείμενο δεν μπορεί να μειώνει την προστασία του καταναλωτή. Και εξού και δυσκολία. Θα σα έδινα παραδείγματα άρθρων που μπορεί να βελτιωθούν αν είχα χρόνο. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε αυτά τα άρθρα, φερειπίν το άρθρο 5, ε, προθεσμία παράδοση, να ε, προσθέσουμε και μία διεύθυνση και ένα τηλέφωνο για τι υπηρεσίε ε, με, μετά την πώληση. Επίση το άρθρο 12, πρόβλημα γιατί μειώνει τα δικαιώματα. Το 46α, το ανέφερε ο κ. Γοσφό, συμφωνώ με την απόψη του και την ανάλυση του, άρθρο 27. περίπλοκο αυτό το μέτρο. Σας παρακαλώ, δώστε μας λίγο χρόνο να συζητήσουμε ένα προς ένα τα άρθρα. Μπορεί να σας φαίνεται ε, δύσκολο κάτι τέτοιο, το να μπούμε σε λεπτομέρειες, να διατάξουμε ολόκληρο κατάλογο με τα άρθρα, αλλά τελικά ο διάβολος κρύβεται στι λεπτομέρειε. Γι' αυτό πρέπει να επισέλθουμε σε αυτές. Κύριε Ζουβέν, συμφωνώ. τμήμα του προβλήματος είναι ότι ποτέ δεν έχουμε χρόνο στι επιτροπέ. Ε, το λάθος το έχουν αυτοί που κανονίζουν τις επιτροπές μας. Αλλά στις 12 Ιουλίου, Δευτέρα, 4 η ώρα, θα έχουμε ακόμα μία ώρα, 45 λεπτά με μία ώρα. Ας είστε εκεί. Τέλο πάντων, τώρα έχουμε το πλήρες συνοποιημένο κείμενο ε, με όλα τα άρθρα και ελπίζω να συζητήσουμε συνολικά τη δομή κτλ. Ούτως ή άλλως, με το στα πλαίσια του ΕΛΚ υπάρχει μια ομάδα εργασία. Ε, Μπορείτε να συνεισφέρετε εκεί για να φτάσετε σε μια κοινή γραμμή. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βαγνιέ. Ο κύριο ε, Χαμπ τον ξαναβάζω στον κατάλογο μιλητών, αλλά η κυρία Βαγνιέ πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να απαντήσω στον κύριο Ζουβεν. Θα μιλήσω με ταπεινοφροσύνη, καταρχήν. Μάλλον είμαι λίγο αμβλήνους για αυτό το θέμα. Γιατί όσο προχωράει η συζήτηση, τόσο μπερδεύομαι και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις ε, κατά, από απόσταση, αυξάνουμε την περιπλοκότητα. Σε επίπεδο υπηρεσιών υπάρχει μεγάλη νομική αβεβαιότητα ακόμα και στο κεφάλαιο 4 φοβάμαι ότι το επίπεδο της προστασίας είναι πιο χαμηλό από τις οδηγίες και εδώ έχω ευρωπαϊκό όραμα και θεώρηση. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε κυρίως τα νέα κράτη-μέλη, όπου η προστασία δεν είναι επαρκής και νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλά πράγματα προς βελτίωση. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε το κείμενο άρθρο προς άρθρο. Παράδειγμα χάρη στο άρθρο 26 ας πούμε. Σημείωσα ότι ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να, ζητήσει τη λύση του, της σύμβασης αν το ελάττωμα συμμόρφωση είναι ίσονο σημασία. Αλλά αυτό εξαρτάται από χιλιάδε πράγματα. Από το επίπεδο προστασία σε κάθε κράτο μέλο. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε σε λεπτομέρειε και να τα ορίσουμε αυτά τα πράγματα. Τα έχω μπερδέψει εντελώ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα και η πρόταση που κάνατε, Πρόεδρε, να έχουμε μια μεθοδολογία, ούτω ώστε να δούμε το σύνολο του κειμένου, όταν έχουμε όλε τι μεταφράσει, με συνεδριάσει και με του ε, θρησκειώδει συζητητέ θα βοηθήσει, γιατί το κείμενο είναι θεμελιώδη σημασία. Ευχαριστώ κύριε Αβανιέ. Κύριο Σάμπατ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το κείμενο αυτό έχω να πω διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι, όπως το είπε και ο Σφαπιάλη νωρίτερα, το διάβημα είναι ένα ενδιαφέρον, ρεαλιστικό διάβημα. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας κύριε Γκέφαρτ, όταν λέτε ότι το σχέδιο του κυρίου Αντρέα Σφάπ είναι ουσιαστικά οπισθοχώρηση σε σχέση με αυτά που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε άλλο και για πολλά σημεία μάλιστα. Έπειτα, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο για το θέμα αυτό να μην έχουμε απλώς και μόνο μία νομική προσέγγιση στο θέμα δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο διασυνοριακό εμπόριο. Και στο κάτω-κάτω η καρδιά της οδηγίας είναι ακριβώ κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και διασυνοριακά του εμπορίου. Οπότε εγώ δεν θέλω να περιοριστούμε στις νομικές πτυχές. Ωραία, πολύ μας αρέσει να βάζουμε νομικά επιχειρήματα, αλλά να δούμε λιγάκι και την οικονομική πτυχή του θέματος. Στόχος μας είναι, πρώτον, η οδηγία αυτή να βελτιώσει οικονομικά και του επιχειρηματίε και του καταναλωτέ. Εγώ θα νομίζω ότι έχουμε από την μια μεριά τους επιχειρηματίε και από την άλλη του καταναλωτέ, Δεν συμφωνώ με αυτή τη στάση. Άρα λοιπόν θέλουμε ανάπτυξη. Αλλιώ γιατί την έχουμε αυτή την οδηγία. Έπειτα, για εμά τουλάχιστον του Γάλλου, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει προστασία χωρί ανάπτυξη. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε την αρμόνιση από μόνη τη Η αναρμόνιση ως αυτό σκοπό, πολύ ωραία. Όμω, δεν είναι αυτό που μα ζητάνε σήμερα οι καταναλωτές. Στη Γαλλία λοιπόν πιστεύουμε ότι την εναρμόνιση, αν θέλουμε να τη βελτιώσουμε, μπορούμε. Είδα ότι υπάρχει το ανώτατο, το ανώτατο συν, το ελάχιστο, τα είδα τα διάφορα άρθρα. Αλλά για τη φιλοσοφία του κειμένου αυτή καθεαυτή πιστεύω ότι η εναρμόνιση δεν πρέπει με τίποτα να μειώσει την προστασία των καταναλωτών. Τώρα πιο συγκεκριμένα στο γαλλικό δίκαιο εμείς έχουμε διάφορες προβληματικές όπως είναι το κρυφό ελάττωμα κλπ. κλπ. Ωραία. Καλά κάνουν και υπάρχουν αυτά στο κείμενο, όμω να μην υπάρχει αβεβαιότητα, να υπάρχει μια ρεαλιστική προσέγγιση, ιδιαίτερα για τι καταχρηστικέ ρήτρε και για άλλα σημεία που δεν προλαβαίνω να σα πω σήμερα. Αλλά το κυριότερο για μα είναι ότι η οδηγία πρέπει να επικεντρώνεται στην καρδιά του θέματο, που είναι η πώληση εξ αποστάσεω. Αυτό δημιουργεί ανάπτυξη. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι σήμερα. Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Είπα ένα λεπτό, ίσως δεν ήσασταν στην αίθουσα. Είχα πει ότι ένα λεπτό ο καθένα έχει στη διάθεσή του. Θα έχετε άλλη φορά την ευκαιρία να μιλήσετε. Δεν ήσασταν εδώ, λέει στα γαλλικά τώρα ο πρόεδρος, όταν είπε ότι ο καθένα σα έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του για να μιλήσει και όχι παραπάνω. Λυπάμαι. Ευχαριστώ, λέει ο μιλητή. Σταματά εδώ λοιπόν. ένα λεπτό να εξηγήσει κανεί όλα αυτά που θέλει για την οδηγία. Ε, δεν μπόρεσα να μπω στι λεπτομέρειε καθόλου. Τι να κάνω. Είναι λίγο το ένα λεπτό. Ένα πράγμα μόνο να πω ακόμα, ότι συμφωνώ με τον σύντροφο πριν που αναφέρθηκε στην προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Πρέπει να έχουμε καιρό να τι μελετήσουμε, τουλάχιστον 20 Σεπτεμβρίου, για να μην πω και αργότερα, τέλη Σεπτεμβρίου, για να ετοιμάσουμε τι τροπολογίε μα. Πρόεδρο, ναι. Λυπάμαι, αλλά έχουμε κι άλλο ένα θέμα. Και γι' αυτό ε, σας έκοψα. Θα πούμε για το χρονοδιάγραμμα μετά. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, ο Μάρτιν Πρόγκ έχει το λόγο και μετά θα επανέλθουμε στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε μια δύσκολη υπόθεση εδώ μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση για συμβιβασμό που έχουμε μπροστά μας. Ακούγοντας τη συζήτηση εδώ σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας τη δομή βέβαια, αλλά να δούμε και τα διάφορα άρθρα αυτά καθε αυτά. Γιατί όταν περνάτε από το ένα θέμα στο άλλο θα δείτε ότι τα δικαιώματα δεν εξαφανίζονται, τουλάχιστον ε, έτσι όπως ε, έχει δικιά μας πρόταση. Αν λοιπόν μεταφέρεται στα κράτη-μέλη την αρμοδιότητα, τα κράτη-μέλη πρέπει να το κάνουν. Αν, όπως προβλέπονταν αρχικά, υπήρχε μια ελάχιστη προστασία, αυτή η ελάχιστη προστασία είναι λογικό να παραμείνει. Μερικές φορές είναι δύσκολο πάντως τεχνικά να φτιαχτεί το κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως έχει να κάνει και διάφορες τεχνικές παρατηρήσεις που αν μου επιτρέπετε θα σας τη στείλω, θα τη στείλω στους εισηγητές και στην γραμματεία όλες μας τις τεχνικές παρατηρήσεις γιατί νομίζω ότι θα σας βοηθήσει στην ε, συνέχιση εξέτασης αυτού του θέματος. Στις δικές μας τεχνικές παρατηρήσεις κυρίως αναφερόμαστε σε σημεία που λείπουν ή σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν αλλά δεν θα μπω τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η βασική ιδέα είναι η ελαστικότητα πρέπει να είναι παρούσα για τα κράτη-μέλη. Παρόλο που η αρχική πρόταση δεν έδινε τόσο πολύ ελαστικότητα, τώρα ναι, αλλά τα εθνικά μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν αποτελεσματική και αναλογική προστασία του καταναλωτή. Να είναι πράγματι προστασία του καταναλωτή, η προστασία αυτή. Και νομίζω ότι ο εισηγητής θα διαλέξει το σύστημα που τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα, αυτή η προστασία. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει, επαναλαμβάνει ότι Έχουμε πολλές προσφυγές από καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν να πετύχουν αυτό που θέλουν μέσω του ίντερνετ, του διαδικτύου, γιατί δεν υπάρχει ο προμηθευτής για νομικούς λόγους. Να σκεφτούμε λοιπόν και αυτό το σημείο για τους καταναλωτές και να ανοίξουμε τους, ε, τις αγορές. Αν το πετύχουμε αυτό, η Επιτροπή πιστεύει ότι θα πετύχουμε μια κατάσταση από την οποία όλοι έχουν να κερδίσουν και οι καταναλωτές και οι παραγωγή συγχρόνως. Ευχαριστούμε κύριε Πρόγκ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή να συνοψίσει που έχουμε φτάσει, να μας επιβεβαιώσει επίσης το χρονοδιάγραμμα και να μας μιλήσει για τη διαδικασία που θέλει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ροσφόρ, La Route είναι μια διαδρομή που ακολουθώ εγώ το καλοκαίρι στις διακοπές μου συνήθως. Να το συμπεριλάβω γιατί νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικό καθήκον για όλους μας. Γιατί τη δομή τώρα. Η δομή ίσως δεν έγινε κατανοητή γιατί στις διαφάνειες παρουσιάζεται όχι η δομή αλλά το τελικό αποτέλεσμα. Είμαι ευγνώμων Μάλκολμ που το ανέφερες. Η δομή είναι ίδια με αυτή που παρουσίασα πριν από τρεις εβδομάδες. Δείτε το κυρία Γκέπχαρτ, έτσι είναι όπως σας το λέω. Οι δύο πρώτες στήλε ήταν τα κεφάλαια 2 και 3 σε πράσινο χρώμα πλήρης εναρμόνιση, 4 και 5 ήταν μικτές πράσινο-κόκκινο. Και σήμερα μίλησα για το δεύτερο μέρος και βλέπετε ότι η δομή παρέμεινε η ίδια, διότι το πρώτο μέρος στην ενοποιημένη μορφή του δεν έχει αλλάξει καθόλου. Το είχατε πάρει και από πριν, παραμένει και σήμερα πήραμε το δεύτερο ε, καινούριο κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να συμπεριλάβω. Μου είπαν ότι θα έπρεπε να λάβω υπόψη μου τις προτάσεις και απόψεις των σκιωδών και των άλλων συναδέλφων και γι' αυτό συμπεριέλαβα και αυτό που είπε η κυρία Τούρνουν και δεν άκουσα κάτι από εσάς κυρία Γκέπχαρτ που δεν το έλαβα υπόψη. Πάντα λαμβάνω υπόψη ό,τι λένε οι συνάδελφοι. Δεν είπα ότι είμαι τέλειος, δεν είπα ότι θα τα κάνω όλα εγώ με ταπεινότητα και με τριοφροσύνη είπα ότι έκανα πολλή δουλειά και σας παρουσιάζω τους καρπούς της δουλειάς, βεβαίως θα καταθέσετε τροπολογίες και βεβαίως ε, είμαι διατεθειμένος να τη συζητήσω μαζί σας. Όμως, και αυτό είναι το πρώτο τελευταίο που θα πω, να είμαστε προσεκτικοί, ούτω ώστε να μην παίρνουν, όπως λένε οι Γάλλοι, φαντάσματα στη συζήτηση. Δεν ε, ε, είχα πρόθεση να καταργήσω το δικαίωμα right to reject, επίσης, για παράδειγμα, υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος της βιομηχανίας που ήρθε και μου είπε γιατί δεν το καταργήσατε, γιατί οι μένοι λένε έτσι, οι άλλοι λένε αλλιώς. Ας δούμε λοιπόν ακριβώς πώς έχει το θέμα. Το ίδιο ισχύει και για τα σε τα κρυμμένα ελαττώματα τα οποία δεν τα πείραξα. Μπορούν να εξακολουθήσουν να υφίστανται όπως και το right to reject. Και αυτό είναι το τελευταίο που θα πω. Αν δεν με τίποτα τότε, γιατί κυρία Τούρνεν, να δούμε το θέμα του ποιο ελέγχει την αναλογικότητα. Ε, τώρα η αναλογικότητα ελέγχεται στα νέα μέτρα, τώρα ελέγχεται και γι' αυτό αναφέρθηκα και εγώ στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που κάνει το σχετικό έλεγχο από τώρα. Και γι' αυτό δεν ε, εισάγω κενά δαιμόνια. Ε, κύριε Ροσφόρη, σας βελτιώσουμε τη διατύπωση. Συμφωνώ απόλυτα να το κάνουμε. Τέλος, Είπα ότι τα έχετε όλα τα έγγραφα, πριν από δύο εβδομάδες πήρατε το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος το πήρατε σήμερα. Έχουμε το, το παραδοσιακό κείμενο στις δύο στήλε που θα το πάρετε το απόγευμα. Δεν μπορέσαμε να προλάβουμε να το μεταφράσουμε και από τώρα σε τρεις μήνες μέχρι και τρεις μήνες θα έχετε όλοι ε, καιρό να τα σκεφτείτε, να υποβάλλετε τροπολογίες, να τις συζητήσουμε και ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες προτάσεις σας. Uh, uh, για το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώνω ότι έχουμε κι άλλη συζήτηση για το θέμα στις 12 Ιουλίου, 4 το απόγευμα μετά την ψηφόφο... μετά ε, τα πρώτα σημεία και θα έχουμε ευκαιρία ε, να ξαναμιλήσουμε όσοι δεν μίλησαν σήμερα, η κυρία Τούρνερ. Για το χρονοδιάγραμμα να πω κάτι. Δεν ξέρω γερμανικά το ενοποιημένο κείμενο λοιπόν εγώ θα το πάρω σε καμιά δυο ή και τρεις εβδομάδες όχι δύο εβδομάδες το νωρίτερο πριν αρχίσουν οι διακοπές. Ναι, αλλά το ενοποιημένο για να συγκρίνεται προς την πρόταση της Κομισιόν Οπότε, σε πραγματικό χρόνο, αν βγάλουμε τις διακοπές, έχουμε στην πραγματικότητα δύο-τρεις εβδομάδες χρόνο γόνιμο για τροπολογίες. Δεν είναι πολύ, μια-δύο εβδομάδες είναι μόνο. Είναι τεράστια η δουλειά, οπότε πρέπει να μιλήσουμε με επιχειρήσεις, με οργανώσεις, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Να προτείνω κάτι. Νομίζω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν, πρέπει να γίνουν απευθείας με τον εισηγητή για τα χρονοδιαγράμματα. Ελπίζω να δεχτεί την πρότασή μου ο εισηγητής. Τώρα που έχετε το πλήρες κείμενο, καλό είναι να συμφωνήσετε μεταξύ σας επί της βασικής δομής της πρότασης, γιατί έτσι η διαδικασία θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα αν συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά, γιατί αλλιώς θα γίνει πολύ περίπλοκο το θέμα, ιδιαίτερα το θέμα της συγχώνευσης κεφαλαίων αν συμφωνήσετε πάνω σε αυτό, καλό είναι. Αλλιώς είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, το ενοποιημένο κείμενο, το λέω αυτό στην κυρία Τούρνεν, είναι πιο εύκολο να παρακολουθηθεί. Όταν αλλάζει ο κύριο Φαπ τις προτάσει τη Κομισιόν, το παρακολουθούμε στο ενοποιημένο καλύτερα από ότι στο δίστηλο κείμενο. Οπότε Μπήκαμε σε μεγάλο κόπο για να φτιάξουμε το ενωπημένο κείμενο και είναι πολύ καλό εργαλείο για τέτοιου είδους περίπλοκες αλλαγές. Οπότε τώρα το έχουμε στη διάθεσή μας όλο το κείμενο με τις ε, αλλαγέ και έχουμε και τις, ε, τη δομή αυτή με τις πολλές στήλε. και ελπίζω ότι στις 12 Ιουλίου που ελπίζω να είσαστε εδώ θα έχουμε ευκαιρία να ε, συζητήσουμε λεπτομερέστερα το θέμα. Ε, κάτι άλλο που ίσως σκεφτούν οι συντονιστές. Έχουμε και 2 Σεπτεμβρίου μια συνεδρία για να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και εκεί εύκολα μπορούμε να προσθέσουμε και συζήτηση πάνω σε αυτό στις 2 Σεπτεμβρίου. Όχι, 13 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, οπότε εντάξει, έχετε χρόνο για συζήτηση. Πάντω εσεί θα τα βρείτε με τον κύριο Σουβάμπ ή Σκιώδη. Κλείνω λοιπόν το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σουάμπ και τώρα θα ήθελα να περάσω σε μια άλλη έκθεση πρωτοβουλίας που αρχίζει σήμερα και θα δώσω την ευκαιρία στην κυρία Χάλτε Μόζερ να το δει για την για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιμένω να περιμένω να ληφθώ μέχρι να βγει ο κόσμος από την αίθουσα. Τέλος πάντων συμφωνήσαμε να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας στην ΙΜΚΟ για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και για θέματα εποπτείας της αγοράς, γιατί υπάρχει σχέση στενή ανάμεσα στα δύο αυτά θέματα. Η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων υιοθετήθηκε το Δεκέμβρη του 2001, εδώ και πολύ καιρό, και θα πρέπει να έχει να έχει εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη από το 2004 και μετά. Η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων έχει γενικές διατάξεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 σκόπευε να κάνει μια αναθεώρηση αυτής της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και έχει οργανώσει ήδη μία διαβούλευση των ενδιαφερομένων για να εντοπιστούν τα ενδεχόμενα προβλήματα αυτής της οδηγίας. Και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας θα πρέπει να αποφανθούμε για το περιεχόμενο της οδηγίας αυτής για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και να πούμε πού πρέπει να ενδυναμώσουμε το κείμενο, πού πρέπει να το αλλάξουμε. Ε, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτή η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων για την οποία μιλάμε σε αυτή την έκθεση. Υπάρχει και ένα άλλο καθεστώς που ρυθμίζει την ασφάλεια των προϊόντων. Θα θυμάστε ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία, στην περασμένη δηλαδή, είχαμε μιλήσει για το νέο νομοθετικό πλαίσιο. που καθορίζει και την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Και ένα πακέτο υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2008 και θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010. Ε, με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουμε την εποπτεία της αγοράς και την καλή γενική ασφάλεια των προϊόντων. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κάποια επικάλυψη ανάμεσα στις διάφορες απαιτήσει, ανάμεσα στις αρχές για την εποπτεία της αγοράς και των υπευθύνων για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Και σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας λοιπόν Θέλουμε να δούμε σε, πρώτο, σε ποιο βαθμό υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο καθεστώτα. Αν υπάρχουν επικαλύψεις, αν υπάρχουν κενά στους κανόνες. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αρχές για την εποπτεία της αγοράς και η παραγωγή έχουν τα πράγματα στο μυαλό τους ξεκάθαρα. Πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι απαιτήσει ε, για τα ασφαλή προϊόντα, γιατί υπάρχουν Εναρμονισμένη τομής, μη εναρμονισμένη τομής που δημιουργούν προβλήματα, αλλά δεν δημιουργούν προβλήματα μόνο αυτές οι διαφορές. Υπάρχει λοιπόν αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και υπάρχουν και οι τομεακές οδηγίες εναρμόνισης. Παραδείγματο χάρη η οδηγία για τα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλοί αριθμοί κανόνες που καθορίζουν εν μέρη την ασφάλεια του προϊόντος και εν μέρη την εποπτεία της αγοράς. Θα διαρωτάστε πώς ε, συνδέονται αυτοί οι κανόνες. Μήπως υπάρχει σύγχυση. Ναι, υπάρχει σύγχυση και φαντάζομαι ότι συγκεχημένα είναι και τα πράγματα στο μυαλό των αρχών για την εποπτεία της αγοράς. Υπάρχουν διάφορα καθεστώτα ε, που εγγυώνται την εφαρμογή των κανόνων. Υπάρχουν καταρχά οι διαφορετικοί νομοθετικοί, διάφοροι μάλλον νομοθετικοί κανόνε. Υπάρχει όμως και μια ιδιάζουσα κατάσταση. Και το φθινόπωρο οι αρχές για την εποπτεία της αγοράς έλαβαν αυτή την έκθεση ε, και προκύπτει από αυτήν ότι κάποιες από τις αρχές δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων. Υπάρχουν πολλοί άριθμοι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς και από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη δεν έχουν επαρκεί πόρου για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Λοιπόν, αυτό το θέμα των πόρων δηλαδή. Επομένω, πώ θα έχω τα πράγματα στο μυαλό μου. Θα πρέπει να εξετάσουμε τρει άξονε, τρία θέματα. Να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ του νέου νομοθετικού πλαισίου και τη οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις απαιτήσει, ε, στους ορισμούς για τους ε, παράγοντες της αγοράς, πώς προσδιορίζουμε τον σοβαρό κίνδυνο στην ε, οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και αν αυτό επηρεάζει την ασφάλεια των προϊόντων. Έχουμε παρκή προστασία στο σύστημα e RAPEX. Ποιες είναι οι απαιτήσει για τις εθνικές αρχές και ούτω καθεξής. Εξετάζουμε λοιπόν τη σχέση μεταξύ του νομοθετικού πλευσίου και τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Εν συνεχεία, σα προτείνω να εξετάσουμε τον κανονισμό για την εποπτεία τη αγορά. αν υπάρχουν περιορισμοί στα κράτη-μέλη που τα εμποδίζουν να εξασφαλίσουν μια καλή εποπτεία τη αγορά, Υπάρχουν οικονομικοί λόγοι που περιορίζεται η εποπτεία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, επαρκείς απαιτήσει για να επαληθεύονται τα προϊόντα. Επαρκεί η νομοθεσία για να είμαστε σίγουροι ότι ελέγχουμε ας πούμε τα προϊόντα που πολλούνται online. Πώς λειτουργεί το καθεστώς ε, εποπτείας της αγοράς. Και τρίτον, η συνεισφορά της ε, συγκεκριμένης οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και μήπως πρέπει να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε τους κανόνες. χάρη για την η χνηλασιμότητα των προϊόντων. Παραδείγματο χάρη, οι Αμερικανοί έχουν υιοθετήσει νέου κανόνε για την χνηλασιμότητα. Τα ακούσαμε πριν από λίγε εβδομάδε σε μία συνεδρίαση. Οι δικοί μα κανόνε για την χνηλασιμότητα είναι επαρκεί. Μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό που συμβαίνει στι ΗΠΑ. Και αν οι κανόνε μα δεν είναι ομοιόμορφοι, ίσω θα πρέπει να ξαναδούμε του κανόνε αυτού χθε κάναμε μία ακρόαση τριών ωρών για την α, τυποποίηση. Υπάρχουν και κανόνε για την τυποποίηση στην α, Οδηγία γενική ασφάλεια των Προϊόντων. Πρέπει να του εξετάσουμε αυτού του κανόνε, αν θέλουμε να έχουμε μία τυποποίηση σοβαρή. Κα... Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Είναι περίπλοκα. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα τις εξετάσουμε αυτές τις απαιτήσει για την τυποποίηση. Κάτι άλλο σημαντικό η νέα διαδικασία για τα επικίνδυνα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Είναι μια νέα διαδικασία που μας δίνει τη δυνατότητα να δράσουμε μέσα στη διάρκεια ενός έτους. Ίσως θα πρέπει να αλλάξει η προθεσμία και να αλλάξει και στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία, απλώς σας λέω κάποια δειγματοληπτικά, ε, για να σας εξηγήσω ότι πραγματικά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Τώρα, πού έχουμε φτάσει μέχρι στιγμή. Ήδη έχω συνεδριάσει μία φορά με τους κοιόδη εισηγητέ. Ζητήσαμε ένα briefing note, ένα ενημερωτικό σημείωμα για κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσα σήμερα. Αυτό το σημείωμα θα το έχουμε ε, στο τέλος Σεπτεμβρίου για τη συνεδρίαση της ΣΥΜΚΟ 29 και 30. Συμφωνήσαμε λοιπόν μεταξύ μα ότι θα οργανώσουμε ένα εργαστήρι και θα σα παρουσιάσουμε αυτό το έγγραφο, το ενημερωτικό σημείωμα. Τότε θα ξέρουμε λίγο περισσότερο πώ έχουν τα πράγματα, ποια είναι τα προβλήματα κτλ. Εν συνεχεία θα παρουσιάσω το σχέδιο έκθεση για να το συζητήσουμε στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ θα έχει μεταφραστεί μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, ας πούμε. Και η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών, προσωρινή, θα είναι αρχές Δεκεμβρίου και φαντάζομαι θα ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ τον Ιανουάριο του 2011 και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου 2011. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, αυτή είναι η διαδικασία που μας περιμένει για αυτό το κείμενο που είναι περίπλοκο, αφορά ένα τεράστιο τομέα. Νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε το απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μας. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχω θέσει πολύ περισσότερα ερωτήματα από ό,τι έχω δώσει απαντήσεις. Ελπίζω να δοθούν απαντήσεις αργότερα και ελπίζω να δώσουμε ένα τελικό κείμενο στην ΙΜΚΟ και ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο τότε μπορούμε να δώσουμε σαφείς υποδείξεις και συστάσεις προς την Κομισιόν που μπορούν να συνεισφέρουν ούτως ώστε να έχουμε ένα καθεστώς εποπτείας αγοράς καλύτερο και να είμαστε σίγουροι ότι η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων είναι μοντέρνα, σίγουρη και αυτό που χρειαζόμαστε. Και ελπίζω λοιπόν ε, να συνεισφέρει η δική μας έκθεση. Περιμένουμε με ανυπομονησία να συνεργαστώ με τους συναδέλφους εφόσον θέλουν να μου παρουσιάσουν ε, χρήσιμες προτάσεις. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εξήγησες με σαφήνεια τη θέση σου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν θέλω να φάμε πολύ χρόνο από τη συνεδρίαση των συντονιστών αλλά όπως είπε και η κυρία Σαλμόζα έχουμε μέχρι τον Ιανουάριο που μας έρχεται, της επόμενης χρονιάς δηλαδή, οπότε δεν επήγει να συζητήσουμε τώρα. Βέβαια οι σκιώδες είναι εδώ, οπότε ίσως θα μπορούσαν να κάνουν κάποια παρατήρηση για τα διάφορα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Ε, αντικαθίσταται κυρία Κορχόλα, σκιώδης εισηγήτρια νομίζω εδώ, από τη συνάδελφο, εκτός αν δεν θέλετε. Θέλετε? Λοιπόν, η κυρία Ρόιτοβα είναι εδώ, εκ μέρους της κυρίας Κορχόλα που είναι σκιώδης, ο κύριος Κρότσμαν, η πράσινη, η κυρία Ρούλε. Και πάλι σκιώδης εισηγήτρια. Και ο κύριος ε, Φόξ, ο κύριος Πενταφυλίδης έφυγε, ο κύριος Αλβίνη δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά σήμερα το πρωί. Έχουμε όμως ο χρόνο στη συνέχεια. Η κυρία Ρόιτοβα λοιπόν πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυρία Καρχολά που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Μου ζήτησε όμως να κάνω κάποια σχόλια εκ μέρου της όσον αφορά την οδηγία αυτή που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των αγορών και την εποπτεία των αγορών. Η εποπτεία της αγοράς, δίχως άλλο, είναι μεγάλη πρόκληση για πολλές χώρες μέλη που δεν καταφέρνουν να βρουν τους σπόρους που θα κάνουν το χείρημα αυτό αποτελεσματικό. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας που θα έπρεπε να κοιτάξουμε προσεκτικά. πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε συνοχή ανάμεσα σε εναρμονισμένα και μη εναρμονισμένα προϊόντα. Έπειτα πρέπει να αναλύσουμε και να δούμε μήπως πρέπει να συνεχίσουμε με τους κανόνες που αποκλίνουν όσον αφορά αυτό το θέμα και αυτό ανάλογα με το τι είδου προϊόντα εξετάζουμε. Έπειτα, οι διαδικασίες ε, τυποποίησης είναι κάτι που πρέπει να δούμε και τις προδιαγραφές πρέπει να τις αναθεωρήσουμε γιατί πολλές φορές ε, οι ρυθμίσεις ε, αργούν πάρα πολύ. Η Επιτροπή λοιπόν θέλει να προχωρήσει ε, συντονίζοντας τις αρμόδιες αρχές στο ερευνητικό στάδιο και σε άλλες δραστηριότητες. Η πρωτοβουλία είναι καλή, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε περισσότερο σε βάθος το εύρος και το κόστος, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσουμε χρήματα από την πραγματική εποπτεία στα κράτη-μέλη. Τώρα, οι γενικέ διατάξει για την ασφάλεια των προϊόντων και τα μέτρα επιβολή είναι πράγματα που επίση πρέπει να δούμε περισσότερο. Τέλο, πρέπει να κοιτάξουμε τους μηχανισμούς που ξεκινάνε να εμφανίζονται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προϊόντα καινούρια που πρέπει να ελεγχθούν για ένα χρόνο και μετά θα έπρεπε η διαδικασία να προχωρήσει. Υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα τα οποία μιλούν για ένα χρόνο και άλλα που λένε ότι πρέπει να είναι πιο μακρά η περίοδος όσο τα προϊόντα θεωρούνται επικίνδυνα. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε πώς θα αποφύγουμε αποκλίνουσες αξιολογήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου τη κυρία Κορχόλα θα της πείτε ότι μας ενημερώσατε. Ο κύριος Κρότσμα είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή πέρασε ο χρόνος, δεν θα βγάλω λόγο. Ε, ήδη αναφέρθηκαν ε, τα προβλήματα από την εισηγήτρια ε, στην εποπτεία της αγοράς στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές αδυναμίες. Στη Γερμανία μίλησα με εκπροσώπους ειδικού από το Υπουργείο Οικονομικών και διαπιστώνουμε ότι όποιος παίρνει στα σοβαρά την εποπτεία, υπάρχουν μερικοί που την παίρνουν στα σοβαρά την εποπτεία, άλλοι όχι. Και είναι σημαντικό εκείνοι που λειτουργούν στην εσωτερική αγορά να εντοπίζουν τις αδυναμίες για να αποφεύγουμε προβλήματα. Γιατί εκεί που υπάρχουν αδυναμίες, εκεί ε, επισημαίνουν και όσοι θέλουν να φέρουν τα προϊόντα τους παρατύπως. Πρέπει να γίνουν λοιπόν συζητήσεις, να δούμε και τι κάνουν οι Αμερικανοί οι οποίοι λέγουν ότι εμείς θέλουμε ανεξάρτητες αρχές να εποπτεύουν την αγορά. Έχουμε το σήμα CE που είναι προαιρετική απόφαση. Υπάρχουν και το CS που δεν ε, είναι καλό, δεν το θέλουν τα κράτη-μέλη όλα, αλλά που όμως δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το κεκτημένο, να έχουμε ελέγχους σωστούς. Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και μάλιστα συζήτησα και έκανα και μία ομιλία για αυτό το θέμα σε ένα ε, ίδρυμα για τους ε, καταναλωτές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Σταματώ εδώ. Πολλά πρέπει να υποθούν, να συζητήσουμε και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική να συνεργαστούμε πάνω σε μια σημαντικότατη έκθεση για την ε, αναεξέλιξη της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ρούλα. Μια λέξη και μία πρόταση. Ε, θα πρέπει να ε, έχουμε μια ε, συμφωνημένη προσέγγιση, να αποφύγουμε τις επικαλύψεις στη νέα προσέγγιση. Τώρα, θα μπορούσαμε αυτή την πρόταση να κάνουμε μια ε, κρόαση για την εποπτεία της αγοράς, γιατί πολλές φορές τα κράτη-μέλη θεωρείται ότι είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν ας πούμε προβλήματα στα παιχνίδια ή στις συσκευασίες ε, και πάντοτε μας ασκείται κριτική ενώ πρόκειται για δυσλειτουργική εποπτεία της αγοράς. Οπότε αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε. Και το θέμα είναι αν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε μια ακρόαση, γιατί το θέμα το θεωρώ πολύ σημαντικό. Θα γίνει εργαστήριο ως αποτέλεσμα της ε, μελέτης. Ο κύριος Πρόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Σάλντε Μόζερ για την πρωτοβουλία της να υποβάλει την έκθεση. Γιατί χωρίς αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς είναι ακαδημαϊκές οι συζητήσεις περί ασφάλειας προϊόντων και επίπεδου νομοθεσίας. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων και όχι να προσθέτουμε συνεχώς νέους κανόνες που σε κάποιες περιοχές της Ένωσης φαίνεται ότι αγνοούνται. Ε, λοιπόν, με μεγάλη χαρά θα σας ε, επικουρήσω στην ε, έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Δεν έχω ζητήσει αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ. Επειδή είστε σκιώδης, είστε μέρος της ομάδας. Σε αυτό το στάδιο καλό είναι να ξέρουμε πώς η Κομισιόν ε, βλέπει όλα αυτά σε σχέση με την αναδιατύπωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Σάλτε Μόζερ και τους Σκιώδης. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι ε, πατήσαμε τα σωστά κουμπιά εδώ. Άρχισε η συζήτηση. Κύριε Φόξ, σας διαβεβαιώνω ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να εισαγάγουμε καινούριου κανόνες. Θέλουμε να εξυγχρονίσουμε την κειμένη νομοθεσία και να φροντίσουμε για καλύτερο συντονισμό για την εφαρμογή. Έχοντα ακούσει και εσά, κύριε Πρόεδρε, πάνω σε όλα αυτά βλέπω ότι συμφωνούμε απόλυτα. Η ουσία του θέματος είναι ε, αν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και η κατάλληλη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Όλα ε, είναι κατάλληλα, θέλουμε να τα βελτιώσουμε, να παλύψουμε παρακλίνουσες ε, ε, προσεγγίσεις και να κάνουμε και έναν εξυγχρονισμό για καλύτερη λειτουργικότητα, χωρίς γραφειοκρατίες, με πιο, να έχουμε πιο ενιαία προσέγγιση και να καλύψουμε και τις αλλαγές στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων. Αυτά προς το παρόν προσθέτω δε ότι είμαστε στην απόλυτη διάθεση του Κοινοβουλίου για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δώσουμε και να πάρουμε ε, συστάσεις, υποδείξεις και γενικά μια συμβολή. Κύριε Μακμίλαν, θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Ναι, όχι. Οι απόψεις σας είναι γνωστές στην Επιτροπή και ούτως ή άλλως όλες οι γνώμες είναι στη διάθεσή μας. Να πω ότι η κυρία Φαρνιό και εγώ και η κυρία Κάμι συμμετείχαμε σε μια εκδήλωση οργανωμένη από την ε, Ισπανική Προεδρία για την Ασφάλεια των Προϊόντων και ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μπορούμε να τα προσθέσουμε και οι συντονιστές θα συζητήσουν την πρόταση ε, να κάνουν και για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων μια εκθέση πρωτοβουλίας. Οπότε μπορεί να υπάρχει συντονισμό μεταξύ των δύο εκθέσεων. Η συγγήτρια για να συνοψίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα τελωνία. Είναι και αυτή μια πτυχή, την οποία εγώ δεν ανέφερα, κακώς το ξέχασα. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Η τυποποίηση και συνδέεται τα τελωνία με την τυποποίηση. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Μπορούμε να αποφεληθούμε λοιπόν ε, από την ε, έκθεση αυτή που θα συντάξουμε για να δούμε τη σημασία όλων αυτών των ε, πραγμάτων για την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές. Αυτά, ευχαριστώ. Είναι μια πρώτη συζήτηση αυτή. Περιμένω τη συνεργασία με όλους σας. Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Λοιπόν, για να συνοψίσω. Θα κάνουμε ε, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου ένα τελιέ θα συμφωνήσουν οι συντονιστές. 11 Οκτωβρίου θα πάει η έκθεσή σας για μετάφραση. Θα το δούμε 26-27 Οκτωβρίου. 6 ε, Δεκεμβρίου ε, για τις τροπολογίες. Φεβρουάριο του 2011 στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε. Αυτά ευχαριστώ λοιπόν που ξεκινήσαμε έτσι τόσο δυναμικά αυτή την πρόταση. Τελείωσε αυτό το τμήμα τη συνεδρίαση. Η τακτική μας συνεδρίαση θα ξαναρχίσει στι 3 η ώρα το απόγευμα. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον καθηγητή Μόντι. Έχουμε όλο το κείμενο της έκθεσής του. Θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις ε, γι' αυτό. Και μετά ε, θα είναι εδώ η κυρία Βάιλερ στις 4 η ώρα για, την για τη μελέτη αντικτύπου αντικτύπου. Α, στο, στην αίθουσα 6Q2. Έτσι, μην αφήσετε καθόλου τα χαρτιά σας εδώ. Δεν θα ξανάρθουμε σε αυτή την αίθουσα. Ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Μόντι στις 3 η ώρα. Και τώρα αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών. Ο,